Now we are ready and then uh, we can start. E Ευχαριστώ συνάδελφοι. Όπως είχαμε αποφασίσει στην συνάντηση των συντονιστών, αποφασίσαμε να οργανώσουμε ένα εργαστήριο εν ώψη των ακροάσεων των επιτρόπων το τμήμα διαμόρφωσης πολιτικής Α οργάνωσε αυτή την ε, συνάντηση, αυτό το εργαστήρι. Θα ξεκινήσω πάρα αυτά γιατί έχουμε και κάποια μικρή καθυστέρηση δίνοντας το λόγο στους εισηγητές μας για να μας παρουσιάσουν τα θέματα που είναι αντικείμενο των ακροάσεων με τους επιτρόπους δίνοντάς μας ένα πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας και υπογραμμίζοντας τα θέματα που είναι κρεμή και για τα οποία θα πρέπει να μιλήσουμε με την Επιτροπή και να συζητήσουμε την Επιτροπή τους επόμενους μήνες και έτη. Το λόγο έχει για την πρώτη παρέμβαση ο κύριος Φίλιπ Σέπελμαν από το Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σε ένα τέταρτο είναι μεγάλη πρόκληση να σας δώσω μια εικόνα της ε, περιβαλλοντικής πολιτικής της Ένωσης και τα εκρεμή θέματα. Θα μπω κατευθείαν λοιπόν στο δικό μου καθήκον δίνοντάς σας μια γενική εικόνα των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η νέα πολιτική περιβάλλοντος, οι παγκόσμιες προκλήσεις, αλλαγή κλίματος που γνωρίζουμε, οι γενικές προκλήσεις, η οικονομική ανάπτυξη συνδέεται με την αύξηση της κατανάλωσης των πόρων και την καταστροφή του περιβάλλοντος. Υπάρχουν και κάποιες προκλήσεις ε, διαθροτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χαμηλή ανάπτυξη, ενεργεία, σημαντική εξάρτηση από πρώτες ύλε εξωτερικού και αλλαγή στο γεωπολιτικό περιβάλλον. Επίσης, εσωτερικά υπάρχει έλλειψη συνοχής ε, στην πολιτική και ενσωμάτωση των διαφόρων πολιτικών σε άλλες, ενώ αναδύεται εμπλοκή μη κυβερνητικών ε, φορέων και μια αύξηση του λεγόμενου soft law. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν αποφάσισε να αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά όντας πρωτοπόρο στην μετάβαση προς τη βιωσιμότητα, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και προωθώντας μια έξυπνη, βιώσιμη και συμπεριληπτική ανάπτυξη. Αυτή είναι η αποστολή της στρατηγικής Ευρώπη 2020 που προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις νέες πραγματικότητες του αιώνα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η περιβαλλοντική πολιτική της Ένωσης βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Αφενός της πολιτικής ανάπτυξης της Ένωσης και των παραδοσιακών μορφών διαμόρφωσης πολιτικής στο περιβάλλον της Ένωσης. Αυτό είναι το ιστορικό πλαίσιο στο με βάση το οποίο πρέπει να, να, να, να αναλύσουμε τα υφιστάμενα ζητήματα. Εδώ έχετε μια γενική εικόνα. Η περιβαλλοντική πολιτική της Ένωσης ανατρέχει σε 40 χρόνια νομοθετικών κειμένων πλέον, θεματικής νομοθεσίας κατά βάση, που αναπτύχθηκε μέσω μια σειρά περιβαλλοντικών προγραμμάτων δράσεως που τώρα αποκορυφώνεται στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για το περιβάλλον και που ακολουθεί την ίδια πορεία θερματική νομοθεσία, αλλά ταυτόχρονα ένα άλλο ένας άλλος δρόμος είναι η πολιτική της Ένωσης για ανάπτυξη μέσω της στρατηγικής 2020 που, που έχει στόχο την έξυπνη και συμπεριληπτική οικονομική ανάπτυξη. Αυτό είναι το πλαίσιο των υφιστάμενων πολιτικών για το περιβάλλον της Ένωσης. Στο 7ο περιβαλλοντικό πρόγραμμα δράσης, PPD, έχουμε την παραδοσιακή θεματική νομοθεσία για το περιβάλλον που θα σας παρουσιάσω και τη νέα υποδιαμόρφωση νομοθεσία που προσπαθεί να ανταποκριθεί στις παγκόσμιες προκλήσεις που προανέφερα και και από την στρατηγική Ευρώπη 2020. Αυτή είναι η κατάσταση. Να σας πω δύο λόγια για το, 5, για το 7ο περιβαλλοντικό πρόγραμμα δράσης. Το ξέρετε νομίζω, καλύπτει μια σειρά θεμάτων υγείας, ένταξης με την στρατηγική Ευρώπη 2020 ενώ διαφυλάσσει και αναπτύσσει το φυσικό κεφάλαιο και αναπτύσσοντας μια οικονομία που είναι αποδοτική στην χρήση πόρων. Resource efficient economy. Αυτό συνδέεται με την οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τις θέσεις εργασίας. Σαφώς ωστόσο το 7ο δέλτα πάει πέρα από την ανάπτυξη και την απασχόληση προσβλέποντας στην ευεξία, στη σωστή και καλή ζωή μέσα στα όρια του πλανήτη μας για υγιείς ανθρώπους. Οι πυλώνες 4I στα αγγλικά είναι η ενημέρωση, σωστή ενημέρωση, στα ελληνικά δεν υπάρχει γιώτα, περισσότερες επενδύσεις, καλύτερη εφαρμογή και μεγαλύτερη ένταξη πολιτικής. Ξαφνικά όμως χάθηκαν οι εικόνες. Κρίμας. Ας μπούμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι της παρουσίασής μου κοιτάζοντας τη θεματική νομοθεσία που έχει διαμορφωθεί την τελευταία 40 ετία, 40 ετία. Για παράδειγμα, ένα από τα ζητήματα που θα αντιμετωπίσετε είναι η νομοθεσία για τον αέρα. Το πακέτο πολιτικής αέρα το νερό, με την οδηγία πλαίσιο για το νερό, υπάρχει σημαντική πρόοδος στον τομέα και θα αναπτυχθεί και εγκριθεί περαιτέρω. Η βιοπικιλότητα, η οδηγία για τους οικοτόπους και για τα πουλιά, για τα πτηνά και η αδυναμία μας να τηρήσουμε τους στόχους της βιο ποικιλομορφίε, όπω είδατε στην ε, επιστολή ανάθεσης αρμοδιοτήτων του κ. Γιούγκερ προσπάθησε να συνδυάσει τι δύο διευθύνσει ενισχύοντα την, ε, τις δύο οδηγίες, συγγνώμη, ενισχύοντα την εφαρμογή του. Αυτό βέβαια είναι ένα συμπέσμα το βίντεο στο 7ο ΠΠΔ, ούτε είναι και σύσταση από πλευρά μα, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα, στην ε, χρήση γης υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα υποβάθμισης του εδάφους με σοβαρές ανησυχίες και κάποια στιγμή θα βρείτε και περισσότερες πληροφορίες για, την για τα παραδοσιακά θεματικά ζητήματα στο κείμενό μας. Πόσο χρόνο έχω. Βασική πρωτοβουλία τώρα για την Ευρώπη 2020 είναι η αποτελεσματικότητα της χρήσης των πόρων. Αυτή είναι μια εμβληματική πρωτοβουλία τη στρατηγική 2020, το κέντρο της στρατηγική για το 2020 και σχετίζεται με το πακέτο κυκλικής οικονομίας. Έχουμε λοιπόν τον οθικό χάρτη για την αποτελεσματική στους πόρους Ευρώπη και ένα πακέτο οικονομίας για την κυκλική οικονομία, ανακύκλωση, αποβλήτων, δημιουργία θέσεων εργασίας και αύξηση της παραγωγικότητας των πόρων βελτιώντα την αγωνιστικότητα της Ένωσης. Αυτό είναι ένα τυπικό παράδειγμα περιβαλλοντικής πολιτικής της Ένωσης του Σταυροδρόμι. Η τρίτη πρόκληση που εντοπίσαμε στο 7ο ΠΠΔ είναι οι βιώσιμες ε, πόλεις ανάπτυξη των πόλεων. Αυτό είναι κάτι, είναι ένα θέμα και της διάσκεψης για τους οικοτόπους ε, το 2016 που αποφασίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη κλασικό παράδειγμα ενοποιημένων ε, πολιτικών για την κάλυψη των προκλήσεων στις μεταφορές, στη στέγαση, των βασικών ανησυχιών δηλαδή των ανθρώπων. Να τους δοθούν απαντήσεις στις ερωτήσεις τους για το πώς μπορούν να ζήσουν καλύτερα στις πόλεις, στον πλανήτη. Αυτές, αυτά είναι τα τρία βασικά θέματα που εντοπίσαμε Α, υπάρχει και η οικολογική ανάπτυξη που είναι ένα από τα βασικά θέματα νομοθεσίας όπου υπάρχει προσπάθεια βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας για να ενισχυθεί η απασχόληση και να δημιουργηθεί η οικονομική ανάπτυξη προωθώντας ή εδώ υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα εργαλείων που μπορούμε να εφαρμόσουμε. Η μακροπρόθεσμη πρόκληση είναι να ενισχύσουμε αυτή τη μορφή καινοτομία με τήρηση όχι μόνο περιβαλλοντικών στόχων αλλά και τους άλλους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι την ανάπτυξη. Κλείνω παρέχοντας σας τα βασικά μηνύματα συνοπτικά. Η περιβαλλοντική πολιτική σήμερα είναι κρίσιμη για να μετατρέψει και να καινοτομήσει στην κοινωνικονομική ανάπτυξη στην Ένωση, παροτρύνοντας και ενθαρρύνοντας την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασία στην Ένωση. Υπάρχουν μια σειρά η υποεξέλιξη θεματικών προκλήσεων που πρέπει να βελτιώσουν την ομοθεσία στου τομεί, τη βιοπικιλότητα, του νερού, του αέρα, της χρήσης γή και των χημικών ουσιών, ενώ υπάρχουν νέα νομοθετικά κείμενα σε τομεί αποτελεσματικότητα ενέργεια, την κυκλική οικονομία, τι πράσινε βιώσιμε πόλει. Αυτή είναι η Γενική Επισκόπηση, Πρόεδρε. Μπορούμε νομίζω να ξεκινήσουμε τις συζητήσεις. Σας ευχαριστώ. Και τώρα να δούμε αν υπάρχουν ερωτήσεις από τους συναδέλφους. Έχετε πρόθεση να θέσετε ερωτήσεις στον εμπειρογνώμονά μας. Πέτερλε. Ευχαριστώ. Για αυτή την εισήγηση. Είμαι πεπισμένος ότι η πολιτική μας στο μέλλον θα είναι πιο επιτυχής εάν καταφέρουμε να εφαρμόσουμε ολοκληρωμένες ε, έννοιες. Ως προς αυτό πιστεύω ότι έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας συζητάμε ιδέες που καλύπτουν πολλούς διαφορετικούς τομείς, οπότε πιστεύω πως χρειάζεται πολλή επικοινωνία ανάμεσα στην ενέργεια, την, ε, ε, την ε, γεωργία και το περιβάλλον. Επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα, κάποια μονάδα για... συγγνώμη, αλλά διακόπτη πρόεδρος, δεν ακούω τα Ιταλικά. Κάποιος λείπει. Κάτι έγινε και δεν ακούει τα Ιταλικά ο πρόεδρος. Κάποιο τεχνικό πρόβλημα. We can try to improve your Italian. Έτσι θα βελτιώσετε και τα Ιταλικά σας. Λοιπόν, ωραία, ε, ε, φτιάχτηκε, ε, μπορείτε να συνεχίσετε. Πιστεύω λοιπόν πως Θα πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσο οι προηγούμενες μας πολιτικές είναι ευθυγραμμισμένες με αυτές τις νέες ολοκληρωμένες έννοιες. Ναι. Εντάξει τα Ιταλικά. Ωραία. Αυτά είχα να πω. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον ε, ομιλητή πώς βλέπετε εσείς, ε, κατά πόσο είμαστε έτοιμοι για αυτή την ολοκληρωμένη ε, τις ολοκληρωμένες αυτές έννοιες. Ναι, ανέφερα προηγουμένως στο πρόγραμμα, για το πρόγραμμα τα τέσσερα α το ένα είναι το integration, η ολοκλήρωση. Πρόκειται για μια πρόκληση που αντιμετωπίζουμε εδώ και καιρό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, τονίστηκε ιδιαίτερα στη διαδικασία του κάρτη που πώς αποκαλείται και αφορά την ανεπαρκή ολοκλήρωση του περιβάλλοντος σε άλλες πολιτικές. Σε αυτή τη φάση τα πράγματα εξακολουθούν να μην είναι απόλυτα ικανοποιητικά και είναι προφανές ότι θα πρέπει να προωθηθεί περαιτέρω η ολοκλήρωση του περιβάλλοντος στις υπόλοιπες πολιτικές. Άλλες ερωτήσεις? Ήθελα να σας ρωτήσω αν θεωρείται θετικά το γεγονός ότι ο Επίτροπός μας θα έχει τρία χαρτοφυλάκια. Και έχει γίνει ολοκλήρωση μεταξύ το ε, θαλάσσιο περιβάλλοντος, αλληλείας ε, και του περιβάλλοντος. Αυτά πιστεύετε ότι έτσι θα ενδυναμωθούν ή θα αποδυναμωθούν. Είναι θετική κίνηση ή κάτι που θα πρέπει να μας ανησυχεί περισσότερο. Well, um, I left my crystal ball at home. Να σας πω κάτι, την ε, μαγική μου σφαίρα δεν την άφησα σπίτι. Δεν μπορώ να σας δώσω επιστημονική άποψη παρά μόνο σε πέντε χρόνια μετά από την εμπειρία που θα έχουμε. Έχουμε εμπειρία σε άλλα κάτι μέλη που υπάρχει αυτό το είδος ε, η συγχώνευση. Ε, όπως στην Αυστρία έχουμε μια μεγάλη ε, συνεργασία για το περιβάλλον, τη γεωργία και τα ύδατα. Και από ό,τι άκουσα μέχρι τώρα είναι ότι οι συνάδελφοι ε, προσπαθούν πάρα πολύ σκληρά και μάλιστα η προσπάθεια αυτή είναι αμφίδρομη. Ε, και άρα θα πρέπει να περιμένουμε ε, βελτίωση των πολιτικών βιωσιμότητας των αλευτικών αποθεμάτων. Από την εμπειρία μου μπορώ να σας πω ότι είναι συνήθως σε θέμα εξουσίας και πολιτικής βούλησης. We have Άλλες ερωτήσεις, όχι. Ωραία, ευχαριστώ τον καθηγητή Φιλιππέ Σέπελμαν. Και δίνουμε το λόγο στον επόμενό μας εμπειρογνώμονο που είναι ο Νίκολας Κρέμπικ από το Ινστιτούτο για το Κλίμα και το Περιβάλλον και την Ενέργεια του Βούπερταλ. Έχετε το λόγο. Um, Όπως γνωρίζουμε όλοι, η κλιματική αλλαγή είναι μια τεράστια πρόκληση. Κολοσιαία θεωρείται μάλιστα από τις μεγαλύτερες που δεν ποτύχει να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα. Αυτά είναι τα κακά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι συνδέεται η κλιματική αλλαγή και με ε, μεγάλες ε, ωφέλειες από τη μείωση της ρήπανσης και από άλλα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής έχουμε μεγάλο ωφέλη για τη δημόσια υγεία. Επίσης, η κλιματική δράση συνδέεται και με μεγαλύτερο πλέον πεδίο τομέων. Έχουμε ε, ε, εντοπίσει τρεις τομείς που είναι για μας βασικοί. Οι διεθνείς ε, διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία για το κλίμα, η στρατηγική και το πλαίσιο για το 2030 για το κλίμα και την ενεργειακή πολιτική και αλληλένδετο με αυτό είναι και η πολιτική για την ενεργειακή απόδοση. Τι γίνεται με τις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Όπως γνωρίζετε αυτό το καιρό διαπραγματευόμαστε μια νέα συμφωνία για το κλίμα η οποία πρόκειται να εγκριθεί του χρόνου στο Παρίσι. Θεωρητικά υπάρχει δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να επαναπροσδιορίσει το ρόλο της ως παγκόσμιος ηγέτης σε αυτά τα θέματα. Μέχρι τώρα οι διαπραγματεύσεις αφήνουν ανάμεικτα συναισθήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει πολύ και πίεσε ήδη για την έγκριση του πρωτοκόλλου του Κιώτο από τότε, αλλά όπως όλοι γνωρίζετε οι διαπραγματεύσεις στην Κοπενχάγη εναβάγησαν. Δεν κατέληξαν ε, στην Παγκόσμια Συμφωνία στην οποία αποσκοπούσαμε το 2009 η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν δεν κατάφερε να δείξει εκεί ηγετική στάση και να οδηγήσει σε επιτυχία τις διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, στο Ντέρμπαν στη συνέχεια κατάφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέσει για ένα νέο είδος συμφωνίας, τοπικά δεσμευτικό, ε, συγγνώμη, νομικά δεσμευτικό, μια ε, εντολή καινούρια. Λοιπόν, είναι ανάμεικτα ε, αποτελέσματα και οι επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεθνώς, τώρα θα πρέπει να δείξει και πάλι ηγετική στάση. Ποια είναι η σημερινή θέση της Ένωσης στα διεθνή τεκτενόμενα. είναι υπέρμαχος μιας ισχυρής διεθνούς συμφωνίας με νομικά δεσμευτικές ε, ρυθμίσεις για όλα τα μέρη, ένα ε, γερό σύστημα για την μέτρηση, την αναφορά και την ε, επαλήθευση της στήρησης των συμφωνηθέντων και ε, τακτική αξιολόγηση των στόχων και των δεσμεύσεων. Ποιοι είναι οι σημερινοί στόχοι και φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί στη δεύτερη περίοδο του πρωτοκόλου Κιώτο να μειώσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κατά 20% και σε σύγκριση με τα επίπεδα του 90 ε, μέχρι το 2020. Εδώ όμως έχουμε πρόβλημα. γιατί σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος 18% έχει μειώσει το 2012 ήδη. Ε, το βλέπετε στην μπλε καμπύλη. Με βάση τα σημερινά μέτρα μπορούμε να πούμε ότι θα μειωθούν και άλλο οι εκπομπές κατά 21% έχουν φτάσει στο 21% το 2020. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, διατηρεί σταθερές τις εκπομπές. Ε, αυτό δεν είναι για μας λίγο φιλόδοξο ε, και καθόλου, τουλάχιστον από πλευρά διεθνών διαπραγματεύσεων και κινδυνεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ να υπονομεύσει την ίδια της την αξιοπιστία που θα έχει αρνητικά αποτελέσματα ως προς τη δική της διαπραγματευτική θέση. Άλλο θέμα είναι ποιος χρηματοδοτεί όλη αυτή την προσπάθεια στην Κανκούν, στις διεθνείς διαπραγματεύσεις τα μέρη συμφώνησαν να κινητοποιήσουν 100 ε, δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως μέχρι το 2020 για να υποστηρίξουν και να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες για να περιορίσει ή να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή. Συστήθηκε λοιπόν ένα πράσινο κλιματικό ταμείο, GCF είναι τα αρχικά στα αγγλικά, ε, που φιλοδοξούσε να είναι πραγματικά η ναυαρχίδα ε, του ΟΗΕ για την ε, κλιματική αλλαγή. Χρειάστηκε πολύ χρόνος να στηθεί αυτό το ταμείο, άρχισε να λειτουργεί φέτο το Μάιο. Τώρα κινητοποιεί κονδύλια, υπάρχει μια τέτοια διαδικασία η οποία ξεκίνησε και έχουν υπάρξει δύο συνεδριάσεις Το Νοέμβριο θα υπάρξει και μια τελική συνεδρίαση όπου θα δεσμευτούν οι δωρητέ με υποσχέσεις χρηματοδότησης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τις διεθνεί ε, διαπραγματεύσεις γιατί θα πρέπει και είναι προαπαιτούμενο για να πετύχει όλη η προσπάθεια να, στο Παρίσι να είναι δεδομένη χρηματοδότηση. Ορισμένα κράτη-μέλη ήδη έχουν δημοσιεύσει τις ε, ε, δεσμεύσεις τους. Στην τελευταία όμως συνεδρίαση στη Βόνη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι δεν είναι πρόθυμη να συνεισφέρει άμεσα στην κεφαλαιοποίηση του Ταμείου. Ε, ξέρετε ότι αυτή τη βδομάδα διεξάγεται σύνοδο κορυφής στη Νέα Υόρκη όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει προθυμία πλέον ε, να συμμετέχει στη χρηματοδότηση. Είναι λίγο σαφή τα πράγματα, λίγο ίξης αφήξης. Αυτό όμως τώρα τι σημαίνει για τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων και την ηγετική στάση που θα τηρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Παρίσι μπορεί να επανέλθει ως πρωταγωνίστρια μεν η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Υπάρχουν όμως κάποια προαπαιτούμενα και βασικά στοιχεία. Πρώτον, να αυξηθεί ο στόχος που είχαμε πριν το 2020 και να ευθυγραμμιστεί με τον στόχο και τη συμφωνία για το 2050. 80 με 95% προβλέπεται μείωση εκεί. Ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι ότι θα πρέπει να δεσμευτούν τα κράτη-μέλη για ένα στόχο μείωσης με τη νέα συμφωνία με την απαραίτητη και κατάλληλη χρηματοδότηση στις αναπτυσσόμενες χώρες για να αντιμετωπίσουν και αυτές την κλιματική αλλαγή και να περιορίσουν τις συνέπειες. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο επίσης είναι ο ρόλος ακριβώς των αναπτυσσομένων χωρών. Οι επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και θετικές και αρνητικές και στη συνεργασία με τις χώρες ε, της αναπτυσσόμενης και η συμφωνία στο Παρίσι νομίζω και όλη η διαδικασία θα εξαρτηθεί και θα κρυφθεί και από αυτό. Χρειάζεται να σφυριλατηθεί μία ε, συμμαχία και πάλι με τις αναπτυσσόμενες χώρες και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Βεβαίως, όλες αυτές οι διεθνείς δεσμεύσεις θα πρέπει να μεταφερθούν σε εθνικές πολιτικές και σε πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το πλαίσιο για το 2030. Στη διαφάνεια που βλέπετε αυτή τη στιγμή περιγράφεται ε, αυτό το δίκτυο και το, το πλαίσιο μάλλον, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, λέει ποιοι είναι οι στόχοι 20-20-20, ε, για το, τη δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια, την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2011 ανέπτυξε και κατήρθησε διάφορες μακροπρόθεσμες στρατηγικές και βάσει αυτών εξέδωσε μια πράσινη βίβλο και ακολούθησαν διαβουλεύσεις. feedback, um, Σε ό,τι αφορά τώρα τις διάφορες θέσεις στην διαβούλευση εκφράστηκαν, ακούστηκε, ήρθε ένα feedback και τελικά αναπτύχθηκε και δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2014 το πλαίσιο για το 2030. Σύντομα να σας παρουσιάσω μόνο κάποιες θέσεις των διαφόρων ε, φορέων. Έχει και θεσμικών οργάνων, έχει σημασία να πούμε ότι η θέση του ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, και αυτά βασίζονται σε επίσημα έγγραφα, ενώ η θέση του Συμβουλίου ε, ε, είναι από ένα σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου που διέρευσε πριν από δύο εβδομάδες στο διαδίκτυο. Άρα δεν είναι επίσημο έγγραφο, απλώς είναι αντανάκλαση από ένα έγγραφο που διέρευσε. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τη μείωση ε, των αερίων του θερμοκηπίου, φαίνεται να συμφωνούν όλοι στο 40% μέχρι το 2030 σε σχέση πάντα με τα επίπεδα του 90%. Συμφωνούν και τα τρία θεσμικά όργανα. Σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες ενέργειες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα στόχο 27%, μη δεσμευτικό ωστόσο, για τα κράτη-μέλη. Εδώ το Κοινοβούλιο λέει ξεκάθαρα όχι. Καταρχάς όχι 27, 30% και να υπάρχουν στόχοι αναχώρα, μεμονωμένοι. Το Συμβούλιο τώρα φέρεται να λέει κάτι ανάμεσα στα δύο. Ναι στο 30, αλλά χωρίς δεσμευτικούς στόχους για τα κρατη Για την ενεργειακή απόδοση. Um, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως στόχο 30% τον Ιούλιο. Πρότεινε αύξηση δηλαδή μετά από πρώτες αρμόδιες υπηρεσίες, Εδώ το κοινοβούλιο ήταν πιο φιλόδοξο και πιο στεναρό στη στάση του. Ε, ζήτησε πολύ ψηλότερο ποσοστό, 40% στόχο και θέλει και με μονομένους ε, εθνικούς στόχους. Το Συμβούλιο με τη σειρά του και πάλι ε, λαμβάνει μια διάμεση θέση και τι λέει, 30% μεν, αλλά χωρίς δεσμευτικούς στόχους για τα κράτη-μέλη. εδώ υπάρχουν περισσότερες διαφωνίες στην ενεργειακή απόδοση. Και αυτή η διαφωνία είναι ανησυχητική γιατί αυτό είναι ο πιο γρήγορος τρόπος και ο πιο οικονομικός να περιοριστεί η εκπομπή των αρίων του θερμοκηπίου. Η ενεργειακή απόδοση λοιπόν. Η στόχοι της Ένωσης είναι μη δεσμευτικοί για το 2020. Εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20% μέχρι το 20% σε σχέση με τις τιμές του 2007 τις βασικές προβολές δηλαδή. Η πρόοδος με την οποία ε, προχωρούμε προς το στόχο αυτό δεν είναι η επιθυμητή και οι τελευταίες αναλύσεις έχουν δείξει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα κάνει οικονομίες στις τάξεις του 19 ή 18,1%. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Εκτός αυτού δεν είναι ότι κάνουμε οικονομίες, είναι ότι έχουμε οικονομική κρίση και έχει μειωθεί η ζήτηση για την ενέργεια. Άρα οι συζητήσεις είναι πολύ σημαντικές για νέους στόχους και διεξάγονται στα πλαίσια ε, του πλαισίου 2030 για τις ενεργειακές πολιτικές. Και το βασικό μήνυμα λοιπόν που πρέπει να βγει από αυτό είναι ότι σύμφωνα με τη θέση του Κοινοβουλίου θα πρέπει να είναι πιο φιλόδοξος ο στόχος και να φτάνει στο 40% για να δώσει κίνητρα για επενδύσεις και οικονομική ανάκαμψη και να μην επανέλθει η ε, κατανάλωση ενέργειας αυτή τη στιγμή ε, βελτιωθούν τα οικονομικά και καταναλώνει ο κόσμος ενέργεια. Επίσης, υπάρχουν προβλήματα στην εφαρμογή της νομοθεσίας και οι επικείμενες αναθεωρήσεις είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Ποια είναι τώρα λοιπόν τα βασικά θέματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να επαναβεβαιωθούν οι στόχοι, να είναι αρκετά φιλόδοξοι και ισχυροί και δεσμευτικοί. Κάθε στόχος είναι τριπλός και ε, θα πρέπει να επιμείνουμε στην πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και που επιθυμεί ένα 40%. Πάντα με σημείο αναφορά στο 2007. Νομίζω σε μια προηγούμενη διαφάνεια είχε πίσω ένα λάθος, ε, έλεγε επίπεδα του 2007 και όχι βασικό σενάριο. Baseline. Όχι, το, το σωστό είναι το baseline, όχι το level. Παρακαλώ να το διορθώσετε αυτό. Ε, επίσης, αυτός ο στόχος του 40% είναι εθνικός και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στην εφαρμογή, διάφορα παραθυράκια που επιτρέπουν ε, ε, να μην εφαρμόζεται σωστά η νομοθεσία και εδώ έχει να διαδραματίσει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για, αυτά όλα είναι προαπαιτούμενα για να είμαστε πάντα ηγέτες σε διεθνές επίπεδο στις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. And now I ask to my colleagues if they have uh, Ερωτήσεις για τον εμπειρογνώμονά μας. Βεβαίω το κλίμα και η ενέργεια είναι, πολύ, είναι αλληλένδετα θέματα. Και αυτό τονίζεται και από το γεγονός ότι θα έχουμε μια χωριστή θέση για την Κομισιόν ε, που καλείται ε, κλιματική δράση και ενέργεια. Και θα ακούσουμε φυσικά στην ακρόαση ε, τον υποψήφιο επίτροπο. Ποια είναι η προσωπική σας όμως γνώμη, θέλω να σας ρωτήσω. Πυρηνική ενέργεια, τι γνώμη έχετε για τη χρήση της μεσοπρόθεσμα, ποια είναι η γνώμη σας. Γιατί νομίζω ότι κυρίως ε, θα πρέπει να τονίσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να τις αναπτύξουμε περισσότερο, ναι σύμφωνο, αλλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές ε, για όσον αφορά την μέσοπρόθεσμη κατάσταση. Η πυρηνική ενέργεια περιγράφεται ως καθαρή μορφή ενέργειας και ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο δημοσιεύθηκε πριν από ε, λίγες μέρες. Έχει γραφτεί από τέσσερις ε, Αμερικανούς ερευνητές και μάλιστα θεωρούν ότι η πυρηνική ενέργεια μπορεί να σώσει τον πλανήτη. Μεσοπρόθεσμα επαναλαμβάνω. Εσάς ποια είναι η δική σας προοπτική προστασία κλίματος και ο βαθμός στον οποίο η ε, πυρηνική ενέργεια μπορεί να θεωρηθεί καθαρή μορφή ενέργειας. Ποια είναι η γνώμη σας και πιστεύετε πως μπορεί να αποτελέσει λύση μέσω πρόθεσμα, όχι πανάκια παντελής, αλλά εν περιπτώσει ένα βήμα προς την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Thank για την πυρηνική ενέργεια, τι να σας πω, δεν μπορώ να δώσω εγώ προσωπικές απόψεις εδώ, αλλά η πυρηνική ενέργεια συνδέεται με τις χαμηλότερες ε, εκκλήσεις ε, αερίων του θερμοκηπίου. Αυτό είναι αλήθεια. Το κόστος και οι κίνδυνοι όμως που συνδέονται με αυτή την τεχνολογία είναι τεράστια, τεράστια και ιδιαίτερα μακροπρόθεσμα. Οπότε Το να τονίσουμε την επάρκεια της ενέργειας, για παράδειγμα, πράγμα το οποίο θα μείωνε βεβαίως σημαντικά την ζήτηση για ενέργεια, ενώ θα αύξανε το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα ήταν ε, πολύ σημαντική στρατηγική. Κατά τη γνώμη μου. Αυτά μπορώ να σας πω. Ευχαριστώ. Thank you very much. And now... Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, εσείς. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ που περιγράψατε κάποια από τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στην Ευρώπη για να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις στο κλίμα. Όμως οι κλιματικές αλλαγές δεν έχουν να κάνουν μόνο με το πώς εκπέμπουμε, εκλείουμε διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Όταν βλέπει κανείς τις κλιματικές αλλαγές και από την άποψη του Επιτρόπου πώς θα αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών, δηλαδή άνοδο στο επίπεδου της θάλασσας, ασφάλεια τροφίμων, ελλείψεις, περίμωση, ε, ε, κινήσεις ε, των λαών, αποψήλωση των όλα όσα συμβαίνουν ως αποτέλεσμα των κλιματικών αλλαγών. Και φοβάμαι πως ε, η οπτική των κλιματικών αλλαγών είναι περιοριστική. Το να ασχολούμαστε δηλαδή μόνο με την εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα και την παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα είναι, είναι σημαντική, σημαντικό αίτιο, αλλά δεν είναι το μόνο. Έχουμε κόσμο στα λάθος μέρη, έχουμε αποψήλωση δασών, έχουμε ρήπανση γενικώ και δεν μπορούμε να μένουμε μόνο σε αυτό το στενό πλαίσιο. Α, ναι, δηλαδή μόλις ε, δει κανείς κλιματικές αλλαγές πηγαίνει το μυαλό του μόνο στο διοξείδιο του άνθρακα. Και επίσης να ρωτήσω την ίδια ερώτηση που έθεσα και στον προηγούμενο μιλητή. Να έχουμε αυτά τα δύο πράγματα που ε, δείχνουν ότι και πάλι έχουμε τις παροπίδες. Και τι μήνυμα στέλνουμε στον κόσμο όταν λέμε ότι σκεφτόμαστε μόνο το διοξείδιο του άνθρακα ενώ θα έπρεπε να βλέπουμε ολόκληρη την εικόνα των κλιματικών αλλαγών και πώς θα μπορέσουμε να σταματήσουμε τα όσα κάνουμε, να τα αλλάξουμε για να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, η αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος δεν είναι μόνο μετριασμό των επιπτώσεων. Η προσαρμογή είναι κομβικού, κομβική σημασία και υπάρχουν πολλές σχετικέ πρωτοβουλίε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ρόλο συντονιστή των δραστηριοτήτων αυτών και σε εθνικό και σε υποεθνικό επίπεδο υποστηρίζοντας την τις τοπικέ κοινότητες να προσαρμοστούν, να αναπτύξουν στρατηγικές, να ανταποκριθούν στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος. Είναι ένα σημαντικό θέμα να μην έχουμε στο μυαλό μόνο το μετριασμό, αλλά και την προσαρμογή και πώς θα αντιμετωπίσουμε δηλαδή τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος και αυτό δεν σχετίζεται μόνο με εσωτερικές πολιτικές της Ένωσης αλλά και προς τα έξω. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα αυξάνονται σε συχνότητα με αρνητικές επιπτώσεις. Η υποστήριξη εδώ είναι κρίσιμη. Ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση. Δεν βλέπω. Ευχαριστούμε τον εμπειρογνώμονα. Προχωρούμε στον επόμενο. Η κυρία Βίντσιαν Κουαντμπάχ, Senior Health Consultant. Παρακαλώ. Καλημέρα θα παρουσιάσω την ενημέρωση για τη δημόσια υγεία. Η υγεία των πολιτών, όπως ξέρετε, είναι αξία της συνθήκης. Ο στόχος της, της Ένωσης είναι να αναπτύξει πολιτική υγεία συμπληρώνοντας τις εθνικές πολιτικές, ενθαρρύνοντας την, τη διακρατική συνεργασία και διευκολύνοντας το συντονισμό. Ο σκοπός λοιπόν της ενημέρωσης για τη δημόσια υγεία είναι να σας δώσω μια επισκόπηση της κατάστασης της δημόσιας υγείας στην Ένωση, τις αλλαγές που εξελίξονται και να περιγράψω πώς θα αντιμετωπιστούν αυτές οι αλλαγές μέσω των θεσμικών ε, πλαισίων της Ένωσης. Θα σας δώσουμε μια εικόνα και συγκεκριμένα εμβληματικά παραδείγματα η γενική εικόνα στον τομέα είναι η εξής. Πρώτον, έχουμε βελτιώσει σημαντικά την υγεία του πληθυσμού στις, ε, στην Ένωση τις τελευταίες δεκαετίες που οδήγησαν στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής. 80,3 έτη κατά μέσο όρο. Υπάρχει καλύτερη πρόσβαση στην υγεία, στην ε, υγειονομική περίθαλψη και καλύτερη ποιότητα. Επίσης αντιμετωπίζουμε δημογραφικές αλλαγές. Υπάρχει χαμηλό επίπεδο γονιμότητας, μείωση σημαντικά ε, των ε, γεννήσεων, ε, του γεννήσεων στην Νότια και Ανατολική Ευρώπη λόγω και της οικονομικής κατάστασης, ενώ έχουμε πληθυσμούς των οποίων η ηλικία αυξάνεται με αύξηση ποσοστών χρονικών ασθενειών ο πληθυσμός των άνω των 65 σαν ποσοστό θα διπλασιαστεί το 2060 και θα υπάρχει και μια αύξηση των νευροεκφυλιστικών ασθενειών όπως το Alzheimer και άλλες ε, μορφές άνοιας. Ο αντίκτυπος ε, της γύρανσης του πληθυσμού θα είναι επίσης η πίεση που θα υποστεί το σύστημα υγείας και πρόνοιας που πρέπει να και προσαρμοστεί για να παρασχεθεί και σωστή περίθαλψη και να είναι βιώσιμο οικονομικά. Μεγάλη πρόκληση. Έχουμε και το θέμα της μετανάστευσης, θετικής μετανάστευσης, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε μετανάστες που έρχονται στην Ένωση και είναι από αυτούς που συμβάλλουν στην αύξηση του πληθυσμού. Εξετάζοντα την οικονομική κρίση και τον αντίκτυπό τη στη δημόσια υγεία, ξέραμε ότι μέχρι το 2008, πριν την κρίση δηλαδή, πριν το ξεκίνημα τη ύφεση, η υγεία ήταν από του ε, ταχύτερου τομεί ε, αύξηση των δημοσίων δαπανών στα περισσότερα κράτη-μέλη, ξεπερνώντα την ανάπτυξη του ΑΕΠ κατά πολύ. Σήμερα με την κρίση, ο προπολογισμό του κλάδου τη υγεία έχει περικοπεί δραματικά στι περισσότερε χώρε τη Ένωση Ιδίω ε, οι δαπάνε που έχουν να κάνουν την προώθηση και την πρόληψη. Βουλγαρία, Εσθονία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ελλάδα, Λετωνία, Ρουμανία, Πορτογαλία και Ισπανία έχουν κάνει τέτοιε περικοπέ. Η έκθεση του ΩΣΑ τον Αύγουστο ε, ανέφερε ότι υπάρχει μια αύξηση στις δαπάνες για την υγεία, αλλά παραμένει χαμηλή στην Ευρώπη. Τα τελευταία λοιπόν χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο εξέτασαν τις επιπτώσεις της κρίσης ε, στην μείωση των προϋπολογισμών υγείας για να δώσουν συγκεκριμένα πλαίσια για την ε, γενοποιημένη δράση. Κατέληξαν ότι οι μειώσεις στον προπολογισμό της υγείας και στα δίκτυα ασφάλειας, η αύξηση της ανεργίας και η φτώχεια είχαν αντίκτυπο στη δημόσια υγεία. Για παράδειγμα, υπάρχει σχέση μεταξύ αύξησης ανεργίας και μικρής αύξη, και αύξησης, αύξησης των ε, ψυχικών διαταραχών. Η μείωση στην πρόληψη μπορεί να έχει και μείζονες επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού κατά συνέπεια έχουμε όλο ένα και περισσότερες ανισότητες ε, στην υγεία και μεταξύ χωρών και εντός χωρών. Είναι σημαντικό λοιπόν για την Ένωση, τον ΠΟΗ και την ΟΣΑ, ε, η επένδυση στην υγεία ως, μείωση, ως τρόπος μείωσης των ανισοτήτων ε, για την συνοχή και την ανάπτυξη έχουν ουσιώδη, έχει ουσιώδη ρόλο. Ποιο, με ποιον τρόπο απαντάει η Ευρώπη στις πολιτικές για την αναγκαιότητα της υγείας. Το 2010 ξεκίνησε η στρατηγική Ευρώπη 2020 για μια έξυπνη και συμπεριληπτική ανάπτυξη. Πρόσφατα, το Φεβρουάριο του 2013, το πακέτο κοινωνικών επενδύσεων έδωσε έμφαση σε στόχους υγείας ιδίω ενισχύοντας τη μεταρρύθμιση των συστημάτων υγείας. Οι στόχοι αυτοί έχουν στόχο τη μείωση κατά βάση των ανισοτήτων στην υγεία, βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα μέσω της υγιούς καινοτομίας, ηλεκτρονική υγεία, Health HTA, ECHI και επενδύοντας σε ανθρώπινο κεφάλαιο, υγεία των εργαζομένων, επενδύοντας και σε προγράμματα υγείας όπως το τα πολιετή προγράμματα υγείας. Πρόσφατα ξεκίνησε το τρίτο πρόγραμμα υγείας για την περίοδο 2014-2020 που έχει σαφείς στόχους που συνδέονται με την πρόληψη την πρόθεση της υγείας, σοβαρούς κινδύνους, πρόσβαση στην ε, περίθαλψη και καινοτομία. Επίσης υπάρχουν και ερευνητικά προγράμματα όπως το Horizon 2020 που ασχολείται με ασθένειες και βελτίωση της έρευνας συγκεκριμένων ε, ασθενειών όπως των εγκεφαλικών. Ποια είναι, ποιες είναι οι προκλήσεις λοιπόν που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πρώτον, αύξηση του βάρους των χρονικών ασθενειών. Δεν μπορούν να γνωριθούν οι χρόνιες ασθένειες, διότι τα στοιχεία σύμφωνα με τον ΠΟΗ, οι τέσσερις βασικές, καρδιαγγειακές, καρκίνους, διαβήτης και χρονικές αναπνευστικές, χρόνιες αναπνευστικές σκοτώνουν ανα τρεις, ε, σε κάθε πέντε ανθρώπους ανά τον κόσμο. Η Ένωση πλήττεται ιδιαίτερα από τις χρόνιες παθήσεις. 77% του συνόλου του βάρους των ασθενειών στην Ευρώπη. Οι χρόνιες ασθένειες είναι υπεύθυνες για το 86% των θανάτων στην Ευρώπη. με δεδομένο αυτό και γνωρίζοντας ότι η γύρανση είναι η βασική παράμετρος της περίθαλψης και υγείας και διότι οι χρόνιες ασθένειες αυξάνονται μεταξύ των νέων γενεών γνωρίζουμε κατά συνέπεια ότι ο ρυθμός των ασθένων που θα έχουν πολλαπλά, πολλαπλές χρόνιες παθήσεις αυξάνεται δημιουργώντας ε, μεγάλη επιβάρυνση στις ασθένειες και αυξάνοντας το κόστος του συστήματος υγείας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν 700 δις ευρώ δαπανώνται στην Ένωση κάθε χρόνο σε χρόνιες παθήσεις που σημαίνει 70% και των ε, συνολικών δαπανών υγείας σε μια χώρα. Οι συγκεκριμένες ασθένειες τώρα, είπαμε καρδιαγγειακές παθήσεις, Καρκίνο που είναι επικεφαλής το 2012 2,6 εκατομμύρια άτομα διαγνώστηκαν με καρκίνο στην Ένωση και 1.260.000 άτομα πέθαναν από καρκίνο ή, επι, ε, επιπλοκές του. η επιβάρυνση εμπολής οφείλεται στον καρκίνο του στήθους του μαστού των πνευμόνων και ο καρκίνος αυτός ο παράγοντας είναι για τον τελευταίο αυτό είναι το κάπνισμα προφανώς. Διαβήτης τώρα. Ε, αυξήθηκε εκθετικά ο αριθμός των ασθενών με διαβήτη τα τελευταία χρόνια. Θα συνεχίσει να αυξάνεται λόγω της ε, αύξησης της παχυσαρκίας μεταξύ όχι μόνο ενηλίκων αλλά και των παιδιών. Χρόνιας, χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις, άσθμα και άλλες ασθένειες επίσης επηρεάζουν. Παράγοντες κινδύνου τώρα. Εδώ μπορεί να γίνει πολλή δουλειά που συνδέονται με τις ασθένειες αυτές. Οι παράγοντες κινδύνου έχουν περιγραφεί και εντοπιστεί επαρκώς από τον ΠΟΗ. Χρήση καπνού, κατανάλωση ενοπνεύματος, ε, μη υγιείς, ε, μη υγιεινές τροφές, ε, έλλειψη άσκησης. Αυτή τη στιγμή 97% των εθνικών προπολογισμών υγείας πηγαίνουν στην θεραπεία. Μόνο 3% καλύπτει μέτρα πρόληψης. Είναι σημαντικό λοιπόν να δουλέψουμε στην προώθηση υγιού τρόπου, ζω... υγιού τρόπου, ζω... υγιούς τρόπου ζωής, ε, διαπίστωση και πρώιμη διάγνωση ασθενειών. Επίσης σημαντικό είναι να δουλέψουμε με, θέματα διαχείρισης ασθενειών, ενσωματώνοντας την ηλεκτρονική υγεία, το e-health, στις παραμέτρους υγείας και στην παράγη παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Μια άλλη πρόκληση μεγάλη ανησυχία για την Ένωση είναι οι μολυσματικές ασθένειες, ιδίω οι νέες απειλές και η αντοχή στην, ε, στα αντιβιωτικά. Προφανώς αυτό στην Ευρώπη είναι λιγότερο τεταμένο από ό,τι αλλού στον κόσμο, παραμένει ωστόσο ένα θέμα λόγω της αύξησης των μολυσματικών ασθενειών στην Ένωση. Φυματίωση με αύξηση του αριθμού ιδίως μεταξύ των μεταναστών, ε, HIV και, άλλες, ε, και άλλα σεξουαλικά μεταδεδομένα νοσήματα, μεταξύ των ευάλωτων ομάδων και των ομάδων κινδύνου ιδίως ε, αυξάνονται τα ποσοστά άνδρες κρατούμενοι ιδίως στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη ένα σημαντικό επίσης θέμα είναι η πατήτης ε, ΣΕ αυξάνεται αυξάνονται τα κρούσματα όλων και περισσότερο μεταξύ των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού που σημαίνει ότι ε, πρέπει να υιοθετηθούν πολιτικές για την αντιμετώπιση αυτών των ε, ασθενειών. Ταυτόχρονα εμφανίζονται νέες ασθενείς ή επανεμφανίζονται παλιές. Η γρήπη H1N1, SARS που είχαμε δει το 2009 και επίσης αυτό που βλέπουμε τώρα ως απειλή είναι η έκρηξη κρουσμάτων του έμπολα αιμορραγική υπηρετή δηλαδή. Η παρακολούθηση και η δημιουργία συστημάτων έγκαιρης περιοδοποίησης για την αντιμετώπιση των πανδημιών είναι κρίσιμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει καθηγητέ γραμμές για αξιολόγηση κινδύνου και, προπαρασ... και, και τιμότητα αντιμετώπισης πολλών ε, ζητημάτων που την κατεύθυνση αυτή. Πολλές ε, κοινέ δράσεις επίσης έχουν αναπτυχθεί για, όπως για τις χρόνες ασθενείς και τον καρκίνο Επίσης έχουμε κάνει κοινέ δράσεις στο AIDS, HIV και τη φυματίωση. Ενώ υπάρχουν και καθοδηγητήριες γραμμές όπως πρωτόκολλα για την ε, αντιμετώπιση της αντιμικροβιακής αντοχής, αφεκτικότητας. Οι σπάνιες ασθένειες ε, είναι επίσης ε, στην κορυφή των δραστηριοτήτων. Κάθε ασθένεια που πλήττει λιγότερο από ένα κατά δύο χιλιάδες ε, πολίτες θεωρείται σπάνια. ωστόσο, ε, το ποσοστό αυτό καλύπτει 27 με 36 εκατομμύρια άτομα. Η δράση της Ένωσης του τομέα είναι πρώτον να καλύψει την έλλειψη συγκεκριμένης ε, πολιτικής υγείας για τις σπάνιες ασθένειες στην Ένωση. Τα τελευταία χρόνια η Ένωση παρότρινε τις χώρες μέλη να υιοθετήσουν προγράμματα δράσης με υποστήριξη του Europlan και ανέπτυξαν ευρωπαϊκά κέντρα αναφοράς, δίκτυα στην ουσία, ευρωπαϊκών κέντρων αναφοράς για να παροτρύνουν τον επιμερισμό εμπειρογνωμοσύνης, να βελτιώσουν την διάγνωση και να βελτιώσουν την ε, περίθαλψη, διότι ε, έγκαιρη διάγνωση και γρήγορη αντιμετώπιση είναι κλειδιά στις ασθένειες αυτές. Η απάντηση λοιπόν της Ένωσης ήταν η κοινή δράση για τις σπάνιες ασθένειες, το Ευρωπαϊκό Κέντρο ε, Αναφοράς για τις σπάνιες ασθένειες, ε, προθεσμία ήταν τέλος του 2013 στην πραγματικότητα και παροχή πιο ευκολότερα προσβάση, πρόσβαση στα φάρμακα. Ξέρετε ότι σε κάποιες χώρες που δεν υπάρχουν που υπάρχει ανάγκη, γρήγορη ανάγκη σε φάρμακα, βελτιώθηκε η πρόσβαση στα φάρμακα αυτά γρήγορα. Άλλες προκλήσεις πολιτικής που έχουν εντοπιστεί για την Ένωση είναι το θέμα της χρήσης ναρκωτικών και της εξάρτησης, στην εξάρτηση είναι βασικό ζήτημα υγείας στην Ένωση, ιδίως για την ε, μετάδοση ε, μολυσματικών ασθενειών, υπατήτηδα, HIV. Επίσης υπάρχει το θέμα της διασυνοριακής ε, περίθαλψης με την σχετική ευρωπαϊκή οδηγία θα ζητήσουμε να, με, με έμφαση στην αντιμετώπιση των ασθενή. Τώρα, η, το e-health, η ηλεκτρονική υγεία, αποτελεί τμήμα λύσεων για βιώσιμη υγεία. υπάρχουν συστήματα, οι περισσότερες χώρες της Ένωσης έχουν ενσωματώσει το e-health στα, συστήματά τους με πιλωτικά προγράμματα, συστήματα ηλεκτρονικής αποζημίωσης κτλ. Σε αυτή τη φάση είμαστε. Ενώ υπάρχουν, υπάρχει το θέμα νέων τεχνολογιών, νέων θεραπείων και, θε, και αντιμετώπισης μιας σειράς ασθενειών που θα αποτελέσει κίνητρα ώστε οι βιομηχανίες να μετατρέψουν αυτά σε προϊόντα για τους ασθενείς. Ευχαριστώ. Ερωτήσεις. Please. Thank you, Chairman. Ja mam kilka pytań do pani eksperta. Zdajemy sobie sprawę, że jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, to ona generalnie Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντως, η προστασία της υγείας είναι κάτι το οποίο αφορά τα κράτη και είναι επιφορτισμένα με την προστασία της. Ε, ωστόσο, νομίζω πως είναι σημαντικό πως η ε, Επιτροπή μας θα πρέπει να ενεργήσει με σοβαρό τρόπο, να τονίσει δηλαδή την πρόληψη. και την θεραπεία. Η υγειονομική περίθαλψη, διασυνοριακές, ε, ε, διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη κτλ. Ταυτόχρονα μαθαίνουμε ότι ένας από τους οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τις ε, νέες ιατρικές τεχνολογίες και τα φάρμακα περνά από τον Επίτροπο Υγείας στον Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς και Επιχειρήσεων ε, και Βιομηχανίας. Γιατί έγινε αυτή η αλλαγή. Είναι προς το συμφέρον της βιομηχανίας ή του ασθενούς. Γιατί οι νέες ιατρικές ε, τεχνολογίες αναπτύσσονται για τους ασθενείς. Πιστεύω πως αυτή η μεταφορά λοιπόν ε, αρμοδιοτήτων δεν είναι λογική. Πριν από λίγα χρόνια είχαμε πάλι το πρόβλημα γιατί ο Επίτροπος Φερχόγγεν που ασχολείται με αυτά τα θέματα και το Υπουργείο Υγείας της Πολωνίας και η Πολωνία ε, είχαμε μεγάλο πρόβλημα διότι, γιατί είχε την εντύπωση ότι υποστήριζε την ε, βιομηχανία αντί για τον ασθενή πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα ότι αυξάνεται το κόστος της θεραπείας διότι τα γενόμενα φάρμακα, γενώσιμα με συγχωρείτε, ε, ε, περιορίστηκαν πάρα πολύ. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν ποια είναι η γνώμη σας από αυτό. Ναι, δύσκολη ερώτηση. Όπως είπα και εξ αρχής, ε, ο ρόλος της Ένωσης είναι μέσω των πολιτικών της να συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές και να εξασφαλίζει ότι θα υπάρχει σωστός συντονισμός και συνεργασία ανάμεσα στις χώρες. Στο συγκεκριμένο θέμα, για τις υπηρεσίες και τα φάρμακα υπήρξε μια κίνηση στην Ένωση ώστε να υπάρξει μεγαλύτερος ρόλος στο συγκεκριμένο η πτυχή. Βεβαίως υπάρχουν και τεράστια οικονομικά συμφέροντα εδώ, αλλά και επειδή ως τμήμα του προγράμματος υγείας 2014 με 20 δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στις σπάνιες ασθένειες, την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη για να μειωθούν οι ανισότητες στην υγεία. Στον τομέα αυτό λοιπόν Η αίσθηση ότι θα έπρεπε να έχουν και αυτή την αρμοδιότητα όσον αφορά δηλαδή τα φάρμακα και τη διαχείριση ήταν αυτοί προσπάθησαν δηλαδή να διευκολύνουν να, να, διευκολύνουν, να δώσουν τη δυνατότητα στις εταιρείες να εμπλακούν στην έρευνα, στην καινοτομία και στο μάρκετινγκ και υπάρχουν διαδικασίες τις οποίες στηρίζει η Ένωση αλλά δεν ξέρω αν μπορώ πραγματικά να απαντήσω στην ερώτησή σας τελικά αν είναι καλό ή κακό που τα φάρμακα δεν είναι μέρος της Ευρωπαϊκής του Ευρωπαϊκού Φαρμακευτικού Οργανισμού, Ιατρικού Οργανισμού. Σε κάποιες χώρες όπως το Βέλγιο τα φάρμακα είναι αντικείμενο μιας, ενός οργανισμού που ασχολείται με τα φάρμακα και τα ε, σκευάσματα, αλλά ξέρουμε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να επιφέρει εδώ μια κοινωνική και οικονομική συνοχή και στον τομέα της υγείας. Ελπίζω να απάντησα στην ερώτησή σας. Thank you. And now, Ευχαριστώ και τώρα η κυρία Μέισνερ και μετά ο Πίτερ. Πέτερ λέει. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Τρεις ερωτήσεις έχω αλλά σύντομα θα τις πω. Πρώτον, η πολιτική υγείας βέβαια παραμένει εθνική πολιτική και τα συστήματα είναι πολύ ε, ε, διαφορετικά και δεν βλέπω στο εγγύς μέλλον ούτε στο απότερο να γίνονται ενιαία. Μεταξύ κρατών μελών, μόνο ανταλλαγή απόψεων μπορεί να υπάρχει ε, για τις διαφορές και τις ε, αποκλήσεις. Το δεύτερο, ε, αναφερθήκατε στο πληθυσμό που γυράσκει και στη μετανάστευση, σωστά, και χρειαζόμαστε και ένα είδος πολιτιστικής φροντίδας, δηλαδή πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι έχουμε περισσότερους ε, μετανάστες στις χώρες μας έχουν άλλη αντίληψη και πολιτιστικά και πολιτισμικά πώς ε, περιθάλπησε έναν ασθενή, τη φροντίδα του δίνεις. Επίσης, επειδή είναι λίγα τα χρήματα, δεν είναι πολλά και για την πρόληψη, έτσι κι αλλιώς, στα κράτη-μέλη, ε, αλλά ήδη υπάρχουν πολλές εταιρείες ιδιωτικές, οι οποίες ασχολούνται πάρα πολύ με πρόληψη και επιχειρήσεις που ενδιαφερόνται όχι μόνο για την υγεία, για τη θεραπεία των εργαζομένων, αλλά και για την πρόληψη υγείας. Μπορείτε να μας τα σχολιάσετε όλα αυτά. Παρακαλώ. Απάντησε. Ναι, ευχαριστώ πρώτα. Για τη μείωση ε, των ανισοτήτων στην υγεία. Υπάρχει ένα ειδικό πρόγραμμα δράσης. Ποια είναι η ιδέα που κρύβεται από πίσω. Να ε, συντονίσουμε ε, οποιασδήποτε δράσεις αποσκοπούν στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των συστημάτων υγείας. Δηλαδή με κοινωνικές πρωτοβολίες, ε, απασχόληση κτλ. κτλ. Για παράδειγμα, μείωση των ανισοτήτων σε προγραμματά που έχουν να κάνουν με την παχυσαρκία βλέπουμε ότι χρόνια νοσήματα πλέον έχουν ε, τα πιο ευάλωτα στρώματα και φτωχά του πληθυσμού και είδαμε και τη συνέπειες οικονομικής κρίσης στη δημόσια υγεία. Ας πούμε, ο κόσμος καπνίζει περισσότερο όταν έχει προβλήματα ανεργίας ή έχουμε περισσότερες ψυχικές διαταραχές κατανάλωση νοπνεύματος σε καιρούς οικονομικής κρίσης. Αυτό προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει μέσω του προγράμματος υγείας 2014-2020. Αυτές τις ευάλωτες ομάδες να τις προστατεύσουμε με στοχευμένες δράσεις, πρόληψη υγείας με δείκτες συγκεκριμένους μετρήσιμους για να μπορούμε να τα αξιολογούμε και όλα αυτά, όλες τις πρωτοβουλίες. Το τελευταίο πρόγραμμα του 2008-2013 κατά της παχυσαρκίας, αυτές οι ε, πρωτοβουλίες έχουν αξιολογηθεί. Έχει γίνει μια ιδιαίτερη προσπάθεια για τη σχολική υγεία ε, με στόχο τα παιδιά και άλλες τέτοιες εμβάλλοντες ομάδες και αυτές ε, οι αξιολογήσεις όλες θα ληφθούν υπόψη στο επόμενο πρόγραμμα για την προγραμματική περίοδο 14 με 20. Ναι, υπάρχουν ανισότητες, υπάρχουν και δείκτες φυσικά και η αξιολόγηση είναι απολύτως απαραίτητη για να μειώσουμε τις ανισότητες. Culture, of course. για τη μετανάστευση και τις πολιτισμικές διαφορές. Στην Ευρώπη παρατηρείται ε, θετική, θετικό ισοζύγιο στην ε, μετανάστευση, αλλά αυτή ξενέρεται και με ε, πανεμφάνιση ασθενειών. Έχει αυξηθεί η φυματίωση, για παράδειγμα. Και είναι πολύ σημαντικό και αυτό το πολιτισμικό στοιχείο που αναφέρατε. Πώς μειώνονται τα περιστατικά με προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας αλλά και προγράμματα ε, διαχείρισης και αντιμετώπισης των ασθενειών. Μιλήσαμε για την ηλεκτρονική υγεία αλλά ε, η ολοκληρωμένη φροντίδα είναι πάρα πολύ σημαντική εκτός από τη θεραπεία Υπάρχουν διάφορα επίπεδα. Έχουμε πρώτα το γενικό γιατρό, μετά τον ειδικό γιατρό, έχουμε κοινωνικούς λειτουργούς. Υπάρχουν πολλοί ε, εργαζόμενοι στην υγεία, το νοσηλευτικό προσωπικό. Πρέπει να συντονίζεται και με πιλωτικά προγράμματα προχωρούμε προς μια πιο ολοκληρωμένη φροντίδα με ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις ομάδες. Πολύ σημαντική είναι η επαγρύπνηση και η παρακολούθηση των ασθενειών για να κάνουμε πάντα πολιτικές με βάση συγκεκριμένα στοιχεία και σωστά μητρώα ε, που να καταγράφουν σωστά στοιχεία. Να στραφούμε πραγματικά στον πληθυσμό που έχει ανάγκη. Ξέρω ότι υπάρχουν χώρες που δεν έχουν καθόλου τέτοια μητρώα. Το Βέλγιο, για παράδειγμα, για τα λιμόδινο σήματα είναι πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση και κατάσταση. Ναι, θα φτιάξουν ένα μητρό. Ας πούμε, δεν έχει το Βέλγιο μητρό για την υπατήτη δεσέ. Πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω το κάλυψα αυτό. Α, για την γύρανση του πληθυσμού. Και πάλι πιστεύω ότι Ε, ακριβώς ε, η γύρανση σημαίνει ότι χρειάζεται και μια φροντίδα παρατεταμένη, αλλά ενιαία και πάλι, γιατί δεν έχει κανείς μόνο ένα νόσημα, ε, ταυτόχρονα μπορεί να είναι ε, πολλές Και τα νοσοκομεία χρειάζονται συνεργασία και συντονισμό. Και οι κλινικοί γιατροί δηλαδή και γενικότερα το νοσηλευτικό προσωπικό και η ηλεκτρονική υγεία έχει εκεί να παίξει τον ρόλο της στις υπηρεσίες υγείας και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Θα πρέπει να είναι πιο συντονισμένες, πιο ενωμένες, πιο συνεργάσιμες για να είναι και πιο αποτελεσματικές τελικά και με λιγότερο κόστος και τα λοιπά. Τελευταία ερώτηση για την καινοτομία και την πρόληψη υγείας τι εννοείται ακριβώς στην καινοτομία. Εννοώ ότι ξέρω στη Γερμανία ε, οι επιχειρήσεις συμμετέχουν ε, στην πρόληψη υγείας. Έχουν ειδικά προγράμματα για τους ε, εργαζομένους, οι εταιρείε για να μην αρρωσταίνουν οι υπάλληλοι. Δεν ξέρω αν υπάρχει καμιά πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων για την πρόληψη υγείας, όχι για τη θεραπεία στη συνέχεια, τα κράτη-μέλη. Uh, um, για παράδειγμα, για την ε, ε διατροφή και τη σωματική άσκηση. Βεβαίως. Υπάρχει μια τέτοια πλατφόρμα, είναι πρόσδεκτες και επιχειρήσεις να συμμετέχουν και ως εταίροι. Βεβαίως μπορούν οι επιχειρήσεις κάλλιστα να αναπτύσσουν προγράμματα πρόληψης για τους εργαζομένους τους. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αυτή η πλατφόρμα για τη διατροφή και την υγιεινή πιο συγκεκριμένα δίαιτα και διατροφή. Βεβαίως και υπάρχουν αυτά τα προγράμματα και αυτή η πλατφόρμα αλλά και η σχολική υγεία μας έχει προβληματίσει πάρα πολύ και εκεί υπάρχουν εταιρείες που συμμετέχουν και σε αυτό το πρόγραμμα. Η Φεραίρο Ρωσέ για παράδειγμα και η Unilever για την προαγωγή της σωματικής άσκησης. Όλο και περισσότερο συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα και, και αυτό καινοτομία δεν είναι γεφυρώνουμε, χτίζουμε γέφυρες μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ενώ μειώνεται όλο και περισσότερο ο κρατικός κορβανάς μπορεί να συμμετέχει η ιδιωτική οικονομία. Γιατί είναι και τμήμα της απάντησης. Ελπίζω να απάντησα στην ερώτησή σας. θα συνεχίσω εγώ να προεδρεύω στη σημερινή μας συνεδρίαση. Ε, ο κύριος Πέτρλε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αυτή τη φορά θα μιλήσω λίγο περισσότερο, γιατί είμαι και Πρόεδρος της ε, Διακομματικής Ομάδας Υγείας αυτό το Intergroup που αφορά ιδιαίτερα τον καρκίνο. Διανύω την τρίτη μου θητεία ως Ευρωβουλευτής και για τρίτη φορά πλέον ακούω αυτά τα πράγματα. Οι στατιστικές είναι κάθε πέρσι και καλύτερα. Δεν βελτιώνεται η κατάσταση, ο καρκίνος κοντεύει να γίνει επιδημία επελάβνη. Ακούσαμε ότι και άλλες ε, αρρώστιες ε, ξαπλώνονται. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και χρόνια τώρα δεν είναι σε θέση να κινητοποιήσουν ε, τα απαραίτητα κονδύλια και να αυξήσουν τις επενδύσεις να φτάσουν στο 3%. Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι η υγεία παίζει σημαντικό ρόλο. Έχουμε μια συνεργασία στην καταπολέμηση του καρκίνου. Μιλούμε για την περίθαλψη, για την πρόληψη και ό,τι άλλο θέλετε. Τελικά όμως οι ασθένειες είτε εμφανίζονται ταχύτερα ή είναι πιο ανθεκτικές τα φάρμακα. Και φοβάμαι ότι θα χάσουμε αυτή τη μάχη με το καρκίνο. Σε λίγο θα είναι οι μισοί Ευρωπαίοι καρκινοπαθείς, ο ένας στους δύο. Κάτι πρέπει να αλλάξουμε στη βασική μας προσέγγιση και θεώρηση. Δεν μιλάω για σύμπτωμα ή συμπτωματική θεραπεία. Θα πρέπει να το δούμε συνολικά το θέμα. Θα επιθυμούσα να κάνουμε μεγαλύτερες προσπάθειες. 28 κράτη-μέλη είμαστε δεν ξέρω διακυβερνητικά πώς θα γίνει αυτό ενωσιακά. Οι πολίτες περιμένουν περισσότερα από μας. Είμαι πεπισμένος ότι θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι για το σύστημα δημόσιας υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλο που είναι και παραμένει βασικά εθνική αρμοδιότητα, το γνωρίζω αυτό, υπάρχουν όλο και περισσότερα πράγματα όμως που μπορούν να λυθούν με επιτυχία μόνο εφόσον συνεργαστούμε σε κοινοτικό επίπεδο. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, θα πρέπει να ε, έχουμε και μια ένωση για την υγεία και όχι διαγωνισμό για τις αρμοδιότητες. Θα πρέπει να μπει και αυτό το στοιχείο της υγείας στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Γιατί αυτή η κρίση στην υγεία θα διαρκέσει πολύ περισσότερο από την κρίση στην οικονομία. Ξέρουμε και το κόστος που αντιμετωπίζουν τα ταμεία, αλλά πρέπει να έχουμε φιλόδοξους στόχου για να προστατεύουμε τον πληθυσμό. Θυμάστε από την εποχή του Επιτρόπου Μπορτ είχε συμφωνήσει να φτάνουν οι επενδύσει στην προληπτική ιατρική στο 5%. Για μένα αυτό είναι βασικό στοιχείο και προϋπόθεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν οπωσδήποτε σε αυτή τη θητεία τουλάχιστον 5%. Έρχομαι τώρα στην ερώτησή μου. Πώς θα ε, αξιολογούσατε το ρόλο της πολιτικής υγείας της Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι τα μεγαλύτερα κενά και ελλείψεις και δεν ξέρω αν ασχολείστε και εσείς προσωπικά με το καθεστώς ε, του κοινού ερευνητικού κέντρου στην Ίσπρια, στην Ιταλία, Ίσπρα, στην Ιταλία. Πώς βλέπετε το ρόλο αυτού του κέντρου εκεί πέρα σε σχέση με τη δημόσια υγεία. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, uh, Ευχαριστώ κύριε Πέτρελε. Έχουμε τρεις επιπλέον ερωτήσεις. Την κυρία Πετιέ, Λόβεν και Φαρία. Προτείνω να ομοδοποιήσουμε τις ερωτήσεις και μετά να δώσουμε το λόγο στην ε, καλεσμένη μας. Ε, έχετε το λόγο λοιπόν. Κυρία Πέτυρ. Ανάπτυξη ειδικών κατευθυντηρίων γραμμών για τα κράτη-μέλη, ε, πράγμα το οποίο θα ε, βοηθήσει τον κόσμο για να έχει καλύτερη υγεία. Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι πολλές φορές σε απομακρυσμένες περιοχές πρέπει να ταξιδέψουν ακόμα και 100 χιλιόμετρα για να φτάσουν στο γιατρό. Δύο γυναίκες την ημέρα πεθαίνουν από καρκίνο του μαστού. Εάν ενεργήσουμε ε, γρήγορα μπορούμε να προλάβουμε αυτή την κατάσταση. Ο κόσμος λοιπόν που ζει στις γεωργικές περιοχές, αγροτικές περιοχές δεν έχει την ίδια πρόσβαση στις ε, υπηρεσίες υγείας, σε εξετάσεις, σε ειδικού γιατρούς, ε, πρέπει να πάψουν αυτές οι διακρίσεις ενώ εκείνοι κάνουν πολλά για μας γιατί εκείνοι παράγουν ε, τις τροφές μας, ε, τη, διατροφή μας και επίσης ε, προστατεύουν το βασικό μας περιβάλλον και μιλάμε για ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Ευχαριστώ η Ιζαμπέλα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Μάλιστα. Θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση Όσον αφορά την μικροβιακή αντίσταση, ε, ε, ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας τον Απρίλιο υπέδειξε αυτήν ως τη μεγαλύτερη απειλή ε, για την ανθρώπινη υγεία, δηλαδή την αύξηση της ανθεκτικότητας των βακτηρίων, των μικροβίων που μπορεί κάποια στιγμή τις αρρώσεις που σήμερα τις ε, θεραπεύουμε εύκολα και γρήγορα να μην μπορούμε να τις ε, αντιμετωπίσουμε πια. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα και μάλιστα φέτος μάθαμε ότι στη Δανία τέσσερις άνθρωποι πέθαναν από βακτήρια τα οποία βρίσκονται ε, κανονικά στα γουρούνια. Πολύ επικίνδυνη κατάσταση που αφορά όλες τις χώρες αλλά και όλους τους τομείς διότι έχει να κάνει τόσο με την υγεία όσο και με τη γεωργία ε, το πώς δηλαδή θα εμποδίσουμε το να καταστεί το θέμα αυτό ένα πραγματικό πρόβλημα. Επίσης γνωρίζουμε ότι στα, στους χείρους στη Δανία αλλά και στις ευρωπαϊκές χώρες εν γέννη 90% των ζώων φέρουν αυτά τα βακτήρια και έχει αυξηθεί η αντίσταση αυτών στα αντιβιωτικά. Η Κομισιόν έχει υπόψη της κάποιο γενικότερο, ευρύτερο, κάποια προσέγγιση στρατηγική για να καταπολεμήσει την ε, ε, τεράστια αυτή απειλή που απειλεί ολόκληρη την ανθρωπότητα θα έλεγα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τελευταία ερώτηση από τον κύριο Φαρία. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η χώρα μας ε, ακολουθεί διαφορετικό δρόμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον ε, ε, δεν κάνουμε τις ίδιες προσπάθειες. Πριν από λίγες μέρες στην Ισπανία ε, ε, αποφασίστηκε το κλείσιμο ενός δημοσίου νοσοκομείου γιατί ε, δέχτηκε να εισάγει έναν ασθενή που υπήρχαν υποψίες ότι είχε τον ιό έμπολα. Ευτυχώς τελικά δεν έγινε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση περιμένει αυτή η επιδημία να έρθει μέχρι εδώ για να ενεργήσει πιο δραστήρια. Σας ευχαριστώ. Και τώρα έχετε την ευκαιρία να απαντήσετε. Yes, so related to the um, first question. Για την πρώτη ερώτηση. Επενδύσεις σε μεγαλύτερη πρόληψη, σε περισσότερη πρόληψη. Να πάμε το 3 στο 5% του προπολογισμού υγείας. και το ερώτημά σας που πρέπει να έχουμε μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Αυτό που κάνει η Ένωση και το είδα και με τα εθνικά προγράμματα καρκίνου και εθνικά προγράμματα σπανίων ασθενειών είναι να θέτεται στόχους. Αν δεν γινόταν κάτι τέτοιο δεν θα είχε κανένα εθνικό πλάνο, άρα μπορούμε να πούμε ότι σήμερα το 2014, οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης έχουν ένα αντικακινικό πρόγραμμα. Όχι ολοκληρωμένο πλήρως, αλλά οι περισσότερες έχουν ένα τέτοιο. Στις σπάνιες ασθένειες υπήρχε η διεθνικό πλάνο. Ο στόχος ήταν ο Δεκέμβριος του σήμερα οι περισσότερες χώρες έχουν ένα εθνικό πλάνο κατά των σπάνιων ασθενειών σε λειτουργία. Πάλι διαφέρει το επίπεδο από χώρα σε χώρα, αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι να θέτει στόχους, είναι σημαντικό. Αλλιώς θα υπήρχαν ακόμα μεγαλύτερες ανισότητες μεταξύ χωρών. Οι χώρες που ανέλαβαν μόνες τους την πρωτοβουλία, άλλες χώρες που ανέλαβαν μόνες την πρωτοβουλία, άλλες όχι. Οι στόχοι αυτοί λοιπόν είναι κρίσιμοι. Το 5% ο ΣΑΠ το λέει χρόνια τώρα ότι ο προϋπολογισμός ε, υγείας για θέματα πρόβλεψης πρέπει να αυξηθεί διότι η θεραπεία είναι πάντα πιο δαπανηρή. Η πρόληψη λοιπόν αποφεύξιμων ασθενειών είναι σαφώς φθηνότερη. Άσε τα άλλα, καπνό, ενόπνευμα, υγιεινή διατροφή, φυσική άσκηση. Αν δουλεύουμε στις παραμέτρους αυτές, αν αλλάξουμε το lifestyle του κόσμου, κερδίζουμε τη μάχη. Προφανώ χρειάζονται πολιτικές στον τομέα αυτό και αυτό δεν είναι εύκολο. Κάθε χώρα έχει προγράμματα πρόληψη. δεν είναι εύκολη διαδικασία, αλλά γιατί να μην θέσουμε στόχο. Βεβαίω. Εξαιρετική θα ήταν η αύξηση του προπολογισμού τη Υγεία. Δεν ξέρω αν απάντησα στην ερώτησή σα Την άλλη ερώτηση για ειδικέ καθοδηγητήρες γραμμές για την ύπεθρο και παρεμβάσει σε πληθυσμό σε απομονωμένες περιοχές. Αυτό θα δημιουργούσε μικρότερες ανισότητες υγείας, γιατί είχα, είπαμε ότι υπάρχει ανισότητα υγείας μεταξύ χωρών και στο εσωτερικό μιας χώρας μεταξύ πόλεων και χωριών υπάρχουν ε, αποκλήσεις. Στην πρόσβαση βέβαια στην περίθαλψη υπάρχουν λιγότερα νοσοκομεία, λιγότεροι γιατροί στο χωριό. Αυτό που αντιμετωπιστεί, αντιμετωπιστεί ιδίω στο επίπεδο της δευτερογενούς πρόληψης, ε, screening ε, και, προ, και έγκαιρη διάγνωση. Η καθυστέρηση στη διάγνωση είναι κακό πράγμα. Οι ασθενείς χρειάζονται καλύτερη ενημέρωση, να αποκτήσουν κυριαρχίες στις αποφάσεις τους, να έχουν πρωτοβουλία, αλλά κυρίως να είναι ενημερωμένοι. Εάν έχουμε αύξηση του καρκίνου του μαστού σημαίνει ότι τα εθνικά προγράμματα πρέπει να δουλεύουν για να παρέχουν συστάσεις και καθηγητήρες γραμμές. Οργανώνοντας ίσως καμπάνιες στην Ήπεθρο για να δώσουν εύκολη πρόσβαση στην υγεία, με αποζημίωση για παράδειγμα σε τέτοιε πρωτοβουλίε. Ξέρουμε, κάποιο το είπε, ότι ο αριθμό των νέων κρουσμάτων καρκίνου, η τεράστια αύξηση των νέων κρουσμάτων καρκίνου είναι ένα θέμα που πρέπει να εξετάσουμε. Θα έδινε λοιπόν προσοχή στις πολιτικές που χρειάζονται να εφαρμόζουν οι χώρες ιδίως για αυτές τις ασθένειες. Τώρα το ερώτημα για την αντιμικροβιοαντίσταση. Μίζον θέμα. Και το έθεσε και ο Πόη που υιοθέτησε καθηγητήριες γραμμές για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών όχι μόνο για φάρμακα, αλλά για πλαίσια περίθαλψης. Όταν λέτε ποια δράση διατομιακή μπορεί να υπάρχει μεταξύ γεωργίας και υγείας για την αντιμετώπιση τέτοιων θεμάτων, θα έλεγα καλύτερα να τα απαντήσει αυτά ο Ρόμπερτ. Τέταρτη ερώτηση. Έμπολα. Και κατά πόσον η Ένωση πρέπει να είναι πιο δραστήρια. Ξέρετε πρόσφατα η Ένωση ζήτησε, α, μάλλον χαρακτήρισε τη, τον έμπολα, σοβαρή παγκόσμια επίγουσα ανάγκη άρα ξεκίνησε σε μια ιστορία αξιολόγησης κινδύνου κτλ, Εξασφαλίζοντα ότι η Ένωση θα ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει την απειλή αυτή. Γνωρίζουμε ότι δεν προστατευόμαστε 100% Ξέρουμε τι γίνεται στην Αφρική. Τα νούμερα που μας δίνουν για την εκθετική αύξηση της ασθένειας μας οδηγεί στο να πούμε ότι πρέπει να είμαστε στο απίκο και να δούμε τι εθνικές μπορούν να δοθούν σε εθνικό επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε πρωτόκολλα υγιεινής, γραμμέ, γραμμές, ε, γρήγορη ενημέρωση για, τους, για τις απειλές, αυτό είναι πολύ σημαντικό και εκεί πρέπει να επενδύσουμε. Νέα απειλή, προφανώς είναι κρίση, παγκόσμια κρίση, η, έννοια, νομίζω, πηγαίνει, η Ένωση πηγαίνει προς σωστή κατεύθυνση. Νομίζω ότι απάντησα. thank you. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πολύτιμη συνεισφορά σας και τις προτάσεις σας στο θέμα αυτό. Και θα προχωρήσουμε τώρα στο επόμενο μέρος του εργαστηρίου μας. Το πάρα πολύ επίκαιρο και σημαντικό θέμα της ασφάλειας των τροφίμων και θα δώσω το λόγο στον επόμενο ομιλητή για να μας κάνει την παρουσίαση, ο κύριος Ρόμπερτ Πέντερσον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα σας μιλήσω για την ε, πολιτική ασφάλεια μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την κατάσταση των πραγμάτων, το ιστορικό υπόβαθρο, σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις. Στη δεκαετία του 80 το θέμα ήταν ε, ε, αμφιλεγόμενο. θα σας παρουσιάσω λίγο το ιστορικό, επαναλαμβάνω, και τις προκλήσεις. Τρεις είναι οι βασικές προκλήσεις διαφορετικές μεταξύ τους, διαφορετικές ε, ήταν και οι διαδικασίες και καταλήγουμε σε αυτές. Ε, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση θα προχωρήσω μέσω στο θέμα. Λοιπόν, τι σημαίνει ασφάλεια τροφίμων και από πού κινούμε και τι κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ο τρόπος και οι πρακτικές που διατηρούμε την ποιότητα των τροφίμων μας, δηλαδή για να μην έχουν ε, μολυσματικούς παράγοντες, μικρόβια κτλ. που μας ε, ε, βλάπτουν στην υγεία μας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιστορικά, ο στόχος ήταν να είναι το υψηλότερο επίπεδο στη δημόσια υγεία, στην προστασία των καταναλωτών, αλλά έχουν τεθεί και ζητήματα όπως είναι και η υγεία των ζώων η αντοχή των μικροβίων στα αντιβιωτικά είναι ένα θαυμάσιο παράδειγμα. Η, η ιδέα ότι η υγεία των ζώων και η υγεία των ανθρώπων είναι αλληλένδετα θέματα. Είναι λίγο ευρύτερη λοιπόν η προοπτική, σε αυτό θέλω να σας μιλήσω και την πολιτική και την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιο είναι το σημαντικό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας το πλαίσιο για την πολιτική ασφάλεια υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, consumer προστασία των καταναλωτών, αλλά και την εσωτερική αγορά. So the... Λοιπόν, Πώς έχει σήμερα η κατάσταση. Υπάρχει η Γενική Νομοθεσία για τα Τρόφιμα το 2002. Η Λευκή Βίβλος που τότε κυκλοφόρησε ήταν ε, μετά από τα μεγάλα διατροφικά σκάνδαλα της σύγχρονης εποχής ε, που ήταν η και εγκεφαλοπάθεια των βοηδών ή άλλος πως οι τρελές αγελάδες. Ε, από εκεί ξεκίνησε η πολιτική της Ένωσης για την ασφάλεια ε, τροφίμων και είναι διαφορετική για το λόγο αυτό από άλλα μέρη του κόσμου. Η αρχή της προφύλαξης η λεγόμενη είναι ένας μηχανισμός ε, που έχει να κάνει με την επιστημονική αβεβαιότητα και το βλέπω έτσι εγώ ως πανεπιστημιακός. Η άλλη προσέγγιση έχει να κάνει με την τροφική αλυσίδα, το σύνολο Δηλαδή, ε, να δούμε ε, όλη την αλυσίδα παραγωγής και πού μπορούν να προκληθούν προβλήματα για την ασφάλεια υγεία. Ε, υγείας και τροφίμων. Στις Ηνωμένες ε, Πολιτείες το βλέπουν αλλιώς χρησιμοποιούν χημικά για ξέπλυμα τροφίμων κλπ. Υπάρχουν κάποια κρίσιμα σημεία και τομείς που πρέπει να αντιμετωπιστούν για να βελτιωθεί η ασφάλεια των τροφίμων. Ε, τμήμα του ιστορικού είναι επίσης αναφορά στο Γενικό Νόμο και τη Λευκή Βίβλο όπως σας είπα. Ήταν εργάσια στη συνέχεια νομοθεσία που σε μεγάλο βαθμό έχει ολοκληρωθεί. Εκκρεμούν κάποια ζητήματα για την ε, υγεία των ζώων ε, και των φυτών η οποία θα ολοκληρωθεί, αναμένεται τουλάχιστον, μέσα στο 14 και το 15. Μην ανησυχείτε, δεν θα χάσετε τη δουλειά σας. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα, δεν τελειώνει η υπόθεση ασφάλειας τροφίμων εδώ. Και ο κανονισμός θα αναθεωρηθεί με βάση τη διαδικασία refit. Δηλαδή να δούμε κατά πόσο η πολιτική μας προσφέρεται για το στόχο που υποτίθεται ότι εξυπηρετεί. Ας πούμε αν υπάρχουν διοικητικέ δαπάνες, ρυθμιστικό κόστος, διοικητικό γραφειοκρατικό άχθος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έχουν παραγγελθεί δύο μελέτες ε, η μία για τη Γενική Νομοθεσία για τα Τρόφιμα και η άλλη για το Σύστημα Εγγύρης Προειδοποίησης. Αξίζει οπωσδήποτε να το συζητήσουμε αυτό και να το μελετήσουμε. Το λέω απλώς ενδεικτικά τώρα. Λοιπόν, αγνοήστε αυτή τη διαφάνεια παρακαλώ απολύτως. Τρεις είναι οι βασικές προκλήσεις εδώ αναφέρονται πολύ περισσότερες. Για να σας δώσω μια ιδέα για τα βασικά και μόνο. Παγκοσμιοποίηση, κλιματική αλλαγή, διμερείς ε, συμφωνίες που αυξάνονται. Το δεύτερο είναι κάποια επίμονα, όπως θα τα χαρακτήριζα, προβλήματα ε, η σαλμονέλα ας πούμε και κάποιες άλλες ε, ε, πάγιες αρρώστιες και, και, βακτήρια που εμφανίζουν αντίσταση στα αντιβιωτικά. Οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται, γενικά μπορεί να είναι προς όφελος της παραγωγής, αλλά υπάρχουν και παρενέργειες που πρέπει να προσέξουμε. Αυτές είναι οι μεγάλες προκλήσεις που θέλω να σας ε, παρουσιάσω με συγκεκριμένα παραδείγματα. Λοιπόν, η παγκοσμιοποίηση και η αλυσίδα παραγωγής και η κλιματική αλλαγή συνδέονται. Το μεγάλο πρόβλημα στην Αμερική είναι ο συνδυασμός κλιματικής αλλαγής και παγκοσμιοποίηση. Έχουμε νέες ασθένειες που έχουν να κάνουν και με τα τρόφιμα και που δεν έχουμε δει στην περιοχή μας στο παρελθόν. Η κλιματική αλλαγή αλλάζει και τους φορείς ε, των μικροβίων, μεταφέρονται με διαφορετικό τρόπο. Ακούσαμε ε, τα παραδείγματα προηγουμένως για νοσήματα που δεν είχαν εμφανιστεί στο παρελθόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. η κλιματική αλλαγή αλλάζει και τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε τα τρόφιμά μας. Έχουμε περισσότερες τοξίνες, κατάλοιπα, ε, εντομοκτώνων, φυτοφαρμάκων. Για να επανέλθω σε αυτά που είπε ο συνάδελφος προηγουμένως. όντως χρειάζεται πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση όταν μιλούμε για την κλιματική αλλαγή, τα συστήματα τροφίμων, ή αλυσίδες τροφίμων κτλ. Στις εμπορικές συμφωνίες φαίνεται όλο και περισσότερο να αυξάνεται η πίεση για ρύθμιση για την ασφάλεια τροφίμων από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η πίεση αυτή νομίζω προέρχεται τόσο από τις κυβερνήσεις που θέλουν να κάνουν τις συμφωνίες ελευθερών συναλλαγών, αλλά και από άλλους φορείς στην κοινωνία και στην ε, παραγωγή τροφίμων. Ορισμένες οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών φοβούνται ότι δεν θα υπάρξει ρύθμιση πριν καταλήξει κάθε φορά η συμφωνία. Υπάρχει ένας φόβος για τις υπερβολικές ρυθμίσεις από Ας πούμε η συμφωνία TTIP, η Διατλαντική Συμφωνία για το Εμπόριο και τις Επενδύσεις, έχει συζητηθεί πολύ εκεί η αρχή της ε, προφύλαξης που είναι κεντρική ιδέα της πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αμφισβητείται αυτό ε, κατά πόσο έχει επιστημονική βάση. Θα επανέλθω στην αρχή της προφύλαξης και στις αβεβαιότητες ε, τις επιστημονικές. Ε, με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Um, λοιπόν, οι παθογόνοι οργανισμοί όπως είναι το καμπυλοβακτηρίδιο και η σαλμονέλα ε, παραμένουν. Και χαίρομαι που αναφερθήκατε στο παράδειγμα από τη Δανία, γιατί ζω στη Δανία και παρόλο που κατάφεραν να εξαλείψουν τη σαλμονέλα, ε, βλέπουμε νέα κρούσματα να εμφανίζονται. Είναι ένα επίμονο πρόβλημα. Δεν το ξεχνάμε. Απλώς τα βακτήρια και τα μικρόβια αναπτύσσουν νέα στελέχη συνεχώς, εξελίσσονται και τελικά εμφανίζουν αντοχή στα αντιβιωτικά και από πλευρά ε, δημόσιας υγείας αλλά και από πλευρά ασφάλειας των τροφίμων είναι τεράστιο αυτό το ζήτημα. Η Μάργαρετ Τσάν από τον, ε, την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας είπε όχι μόνο ε, περνάμε σε έναν κόσμο χωρίς αντιβιωτικά αλλά στον κόσμο μετά τα αντιβιωτικά. Ε, λοιμώδεις νόσους που αντιμετωπίζαμε στο παρελθόν δεν θα μπορούμε να τις αντιμετωπίζουμε με ευκολία. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Γιατί μια γρατζουνιά στο γόνατο ή όταν πονάει ο λαιμό σα μπορεί να γίνει μοιραίο να αποβεί, πάρα πολύ επικίνδυνο. Αυτά για την ασφάλεια των τροφίμων. Πώς συνδέεται όμως αυτό με τα τρόφιμα, γιατί ακριβώς η αντοχή στα αντιβιωτικά των μικροβίων συνδέεται ε, με τα συστήματα ε, παραγωγής και εκτροφής των ζώων. Και η αντοχή στα αντιβιωτικά έχει να κάνει όχι μόνο με την εντατική κτηνοτροφία, ε, αλλά και με την πυκνότητα των ζώων στο χώρο εκτροφής. Και επίσης αυτό έχει να κάνει και με τη ζωοτεχνία, δηλαδή τη διασταύρωση και την αναπαραγωγή των ζώων. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει και την Επιτροπή σας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι διατομιακό, είναι ένα θέμα συνεργασίας ε, γιατρών ε, ασχολουμένων με τη γεωργία και με το περιβάλλον. Ίσως χρειάζεται κάπως πιο συστηματική προσέγγιση στον τρόπο που γίνεται. Μπορεί να γίνεται ήδη. Το επόμενο παράδειγμα για την αρχή της ε, προφύλαξης είναι το εξής. Ένα από τα πράγματα που θα έχετε να αντιμετωπίσετε στη θητεία σας είναι οι ουσίες που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μόλις ένα οδικό χάρτη για το πώς θα εκπονηθεί μια στρατηγική κατά αυτών των ουσιών. Τι είναι αυτές οι ουσίες. Πολύ σύντομα να εξηγήσω, δεν θέλω να μπω σε πάρα πολύ τεχνικά και λεπτομέρειες. Είναι ουσίες που αναστατώνουν τις ορμόνες μας και τις λειτουργίες του οργανισμού, επεμβαίνουν στο ενδοκρινικό σύστημα και το ε, ε, διαταράσουν και έχουμε προβλήματα από προβλήματα αναπαραγωγής, ε, στηρότητας μέχρι και καρκίνο που συνδέεται με το ενδοκρινικό παθήσεις των αδένων και όλο και περισσότερο παχυσαρκία ή υπερβολικό βάρος. Κανονικά η διαχείριση του κινδύνου τι σημαίνει. Με αυτές τις ουσίες δεν λειτουργεί πολύ καλά, διότι όταν προσπαθούμε να ορίσουμε κάποιες τιμές, δεν φταίει η δόση για την ουσία που προκαλεί ε, την ενδοκρινική διαταραχή, αλλά η διάρκεια ε, της έκθεσης. Δηλαδή δεν είναι πόση δόση παίρνεις, αλλά πόσο χρόνο εκτίθεσαι σε αυτή την ουσία που προκαλεί ορμονικές διαταραχές. Γι' αυτό η αρχή της προφύλαξης εντάχθηκε στην πολιτική ασφάλεια τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί μας δίνει ένα δρόμο για να νομοθετούμε σε τομείς που υπάρχει και επιστημονική ανασφάλεια καμιά φορά. Ξέρετε ότι τα δύο μεγάλα στοιχεία ε, στην ευρωπαϊκή πολιτική ήταν αυτή η αρχή της προφύλαξης και η παρακολούθηση όλης της τροφικής αλυσίδας. Η μίλησε για τις διαπραγματεύσεις και πώς αυτές επηρεάζονται από τις πιέσεις. Ωραία. Τελευταίο παράδειγμα που θέλω να σας δώσω είναι ο ρόλος της τεχνολογίας. Βιοτεχνολογία, νανοτεχνολογία, γενετική τροποποίηση τροφίμων και ζωοτροφών μας έφεραν αντιμέτωπους με μεγάλες προκλήσεις και νομοθετικές νομίζω στο μέλλον θα τις βρούμε μπροστά μας. Ε, τα μεταλλαγμένα είτε είναι τροφές είτε είναι ζωοτροφές ε, είναι ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ και τη λήψη των αποφάσεων γιατί τώρα τι συμβαίνει ουσιαστικά. Έχουμε μια επανεθνικοποίηση του δικαιώματος απαγόρευσης καλλιέργειας ε, μεταλλαγμένων τροφίμων ή ζωοτροφών. Και πάλι επικρατεί εκεί μια βεβαιότητα, η ανασφάλεια επιστημονική και οι αποφάσεις συχνά ε, μπορεί να βασίζονται σε μία μη επιστημονική μέθοδο. Υπάρχουν προκαταλήψεις, αλλά υπάρχουν και ε, στα στοιχεία που προβάλλονται και πρέπει να έχουμε μία προσέγγιση συστηματική ε, που να μελετάει την διάδραση μεταξύ συστημάτων παραγωγής, ανθρώπων και οικοσυστημάτων. Όλα αυτά μαζί. η επιστήμη πολύπεται όταν συζητούμε για τέτοια περίπλοκα ζητήματα και αλληλεπιδράσεις. Ως προς την νανοτεχνολογία τώρα, και είναι το τελευταίο που θέλω να αναφέρω, αυτή μπορεί να είναι μέρη ωφέλιμη, αλλά χρειάζεται πάρα πολύ προσεκτικά να κοιτάξουμε ε, αν είναι περισσότερα τα ωφέλη ή οι ζημίες. Τι εννοώ. Ας πούμε η κλωνοποίηση των ζώων που δεν το έχω βάλει στην παρουσίασή μου και η ανατεχνολογία. είναι ζητήματα που εξετάζονται και τα δύο από τη νομοθεσία περί νέων ε, τροφίμων. Novel food. Η κλωνοποίηση έχει να κάνει με στοιχεία δεοντολογικά και ηθικά, ενώ η νανοτεχνολογία είναι πολύ πιο περίπλοκο. Και δεν είμαι βέβαιος ότι η τεχνολογία των νέων τροφίμων και η αντίστοιχη νομοθεσία μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα περίπλοκα όσο και ευρέα ζητήματα. Η νανοτεχνολογία μπορεί να βελτιώσει τη ζωή μας βέβαια, αλλά μπορεί να έχει και αρνητική επίδραση σε σχέση με το περιβάλλον, τη δημόσια και την ασφάλεια γενικά υγείας. Λοιπόν, εδώ τελειώνει η παρουσίασή μου. Με χαρά να απαντήσω σε ερωτήσεις. Έχω κάνει και εγώ μια ερώτηση εδώ. Και είναι από τα μεγάλα ερωτήματα πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με την πολιτική της να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στην υγεία των τροφίμων και να βρει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Εδώ το ερώτημα λοιπόν και μεγάλη πρόκληση. Η ασφάλεια τροφίμων πιστεύω ότι είναι ένα τμήμα μόνο μια ευρύτερη πολιτική για τα τρόφιμα και πιστεύω ότι θα πρέπει να μας προβληματίσει αυτή η περιπλοκότητα. Ασφάλεια τροφίμων, δημόσια υγεία, κοινωνικοί παράγοντες, διατροφή, ε, νοσήματα που συνδέονται με τη διατροφή. Έχει επικεντρωθεί πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το θέμα, αλλά μήπως να το δούμε πιο συστηματικά, όχι μόνο στενά την ασφάλεια τροφίμων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι όλοι μας προσπαθούμε να βρούμε απάντηση στα ερωτήματά σας. Ισορροπία μεταξύ επιχειρήσεων και υγείας και περιβάλλοντος. Έχουμε και στο παρελθόν καλές σχετικές εμπειρίες. Ανοίγω το Λόγω για συζητήσει. Ο κύριος Στάς. Κάποιος άλλος. Υπάρχουν ερωτήσεις. Θα μαζέψουμε τις τέσσερις ερωτήσεις. Και ο κύριος Πέντεσον θα απαντήσει. Μπάρτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις έχω βασικά. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πέντερσον. Πάρα πολύ καλή η παρουσίασή του και πολύ συγκεκριμένη και απτή. Παρουσίασε πολύ ωραία και σκιαγράφησε τις προκλήσεις. Δύο ερωτήσεις. Μια μικρή για το TTIP, τη Συμφωνία για τις Επενδύσεις με τις Ηνωμένες και το εμπόριο. Και μπορεί αυτό να σημαίνει κινδύνους και απειλές για τη δική μας ασφάλεια τροφίμων και την ομοθεσία μας. Και εσείς ο ίδιος το είπατε για την αρχή της προφύλαξης και αυτή μήπως θα μπορούσατε λίγο να επεκταθείτε όμως την απάντησή σας. Με ποιο τρόπο δηλαδή μια τέτοια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου και πολύ συγκεκριμένα ε, μπορεί να επηρεάσει κάποια κεφάλαια της νομοθεσίας μας για την ασφάλεια τροφίμων. Η πάντα και στις εντολές των επιτρόπων υπερασπίζεται τον εαυτό της και λέει «Καλά δεν θα επιτρέψουμε κρέας με ορμόνες». Ε, ούτε μεταλλαγμένα και τέτοια πράγματα. Εντάξει, είμαστε υπέρ των πιο αυστηρών προδιαγραφών, αλλά τι γίνεται με τη συμφωνία τίτη, πώς επηρεάζει και αν επηρεάζει την νομοθεσία μας. Και δεύτερη ερώτηση, για τα μεταλλαγμένα, τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Το Mission λέτε ε, προς τους επιτρόπους που έστειλε ο κύριος Γιούνκερ για την αποστολή τους λέει ότι εντός εξαμήνου ε, ε, θέλει να αλλάξει η νομοθεσία για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Γιατί το είπα αυτό τώρα, τζάμπα δήλωση είναι, δεν ήταν υποχρεωμένος να το κάνει. Ε, ε, το είπατε κι εσείς, πρόκειται περισσότερο για επανεθνικοποίηση των αποφάσεων ε, για τα γενετικά τροποποιημένα. Υπάρχει τώρα μια πρόταση η οποία είναι ένας μοχλός, μια, ένα μέσο πίεσης έτσι ε, ώστε ε, να προχωρήσει η νομοθεσία. που έχει τώρα οδηγηθεί σε εμπλοκή ε, στο Συμβούλιο διότι δεν υπάρχει δική πλειοψηφία ούτε προς τη μία ούτε προς την άλλη κατεύθυνση. Και τώρα θέλουν να το υπερψηφίσουν στο Συμβούλιο αλλά μπορούν με κάποιες παρακάμψεις που το επιτρέπουν να συνεχίσουν να το απαγορεύουν για τους κατοίκους των χωρών τους. Το πιο επιθυμητό θα ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση να φέρει μία πρόταση για να γίνει πιο δημοκρατικός ο τρόπος λήψης αποφάσεων στο Συμβούλιο. Και αν πραγματικά, και όντως υπάρχει μια πλειοψηφία των κρατών που είναι κατά της έγκρισης ε, των μεταλλαγμένων αυτών, να περάσει η νομοθεσία. Μπορείτε να μας το σχολιάσετε αυτό, παρακαλώ. Uh, Επόμενη ερώτηση, Πύρχα. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μας φοβήσατε για τις προκλήσεις του μέλλοντος, ε, κύριε Σιγητά. Εγώ μιλάω όμως για την αυριανή, μεθαυριανή ακρόαση. Έχουμε πολύ αυστηρούς κανόνες, αλλά στην πράξη δεν γίνεται τίποτα για την ασφάλεια υγείας στην Ευρώπη. Ο Guardian πριν από λίγους μήνες, αλλά και, άλλες, ε, και άλλα δημοσιεύματα στις ΕΙΠΑ, ανέφεραν ότι τα δύο τρίτα των ε, πουλερικών στα καταστήματα στη, στον κόσμο έχουν ε, μολυνθεί από ε, καμπυλοβακτηρίδια. Ε, η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου Ένωσης είπα προβλέπει ότι θα υπάρχει ελευθερία κυκλοφορίας για τα προϊόντα αυτά. Τι σημαίνει αυτό, θα γεμίσουμε ε, με κοτόπουλα αμερικάνικα, με, τέτοιες, ε, με τέτοιους κινδύνους. Αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν τώρα. Κάτι άλλο. Ο κανονισμός του επίπεδου του ύψους ορμονικής παρουσίας. Δεν υπάρχουν διαδικασίες η αλλαγή της νομοθεσίας σημαίνει ότι στην παραγωγή κρέατος, βόλιο κυρίως, η χρήση ορμονών είναι σύνηθης, διότι αυξάνει την ανάπτυξη του ζώου. Άλλο ε, σοβαρό θέμα, για τη μικροβιακή ανθεκτικότητα υπάρχει αύξηση σε στην αντοχή σε αντιμικροβιακές ουσίες. Τα τελευταία χρόνια δεν δημιουργήθηκε κανένα νέο αντιβιωτικό που να αντιμετωπίζει το ζήτημα. Τελευταίο ερώτημα. Το εμπάργο στην Ρωσία. Το εμπάργο της Ρωσίας που προκύπτει από αδύναμες ρυθμίσει στην Ένωση για την ε, ε, μόλυνση των τροφίμων. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για το εμπάργκο. Ξέρετε καταρχάς την κατάσταση. Ο κύριος Μπάλτσου. Ευχαριστώ πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Κύριε Πίτερσον, Μιλήσατε στην δήλωσή σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πολιτική ασφάλεια φήμων. Είπατε ότι περιέχονται πολλά θετικά στοιχεία πολιτικής. Μια πολιτική από το αγρόκτημα μέχρι το πιάτο. Η αφετηρία μας είναι προφανώς να εξετάσουμε όμως τι παράγουμε. Αυτή τη στιγμή Ένα σημαντικό θέμα για την επιτροπή μας είναι οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, ο περιορισμός ή η απαγόρευση των οργανισμών αυτών από τα κράτη-μέλη. Ποια είναι η άποψή σας, μπορεί να απλοποιώ τα πράγματα, αλλά θέλω να ξέρω από πού ξεκινάμε την ελευθερία κυκλοφορία στο πλαίσιο της κοινής αγορά, της ενιαίας αγοράς και τις επιπτώσεις που σημαίνει τι πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη, να μαζεύουν, ε, να συλλέγουν δεδομένα και να εξετάζουν αν μπορούν να επιβάλλουν απαγόρευση σε γενετικά τροποποιημένου οργανισμού σε μια ενιαία αγορά ή μήπως δείτε το από άλλη πλευρά η αφετηρία μας θα πρέπει να είναι η προστασία του περιβαλλοντο να εξασφαλίσουμε δηλαδή ότι ο πληθυσμός προστατεύεται αν ναι ποιες περιστάσεις επιτρέπουν την άρση της απαγόρευσης των γενικά τροποποιημένων. Με άλλα λόγια, ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να επιτρέψει γενικά τροποποιημένα προϊόντα. Πώς μπορεί να το κάνει στο πλαίσιο μιας ενιαίας αγοράς. Θα είναι δημοκρατική αυτή η απόφαση. Καλαμπόκι. Στο Συμβούλιο 28 κράτη μέλη υπάρχουν, εκ των οποίων τα 19 είπαν όχι, 5 είπαν ναι και 4 πήχαν. Υπήρχαν λοιπόν 19 κατά και 5 υπέρ, αλλά αυτό δεν ήταν επαρκές και η απόφαση επανήλθε στην Επιτροπή, τουλάχιστον αυτό κατάλαβα εγώ. Τι άποψη έχετε γι' αυτό. Ο κύριος Πέτερλε. Ευχαριστώ. Δεν έχω να κάνω ερώτηση. Σχόλια θα κάνω. Η λύση καταρχάς είναι να θέσουμε μπροστά του καταναλωτή, νομίζω το ξέρουμε αυτό όλοι, αλλά όταν λέμε για την εξορρόπηση διαφόρων συμφερόντων, μπορεί ο καταναλωτής να μην είναι στο κέντρο της προσοχής. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, αλλά δεν είναι πάντα η αλήθεια της πλειοψηφίας. Ως καταναλωτής, αν είμαι πεπισμένος ότι κάτι είναι επιβλαβές, δεν θέλω να διαπραγματευθώ, δεν θέλω να το συζητήσω. Αυτό έτσι βιώνουν πολλά πράγματα οι καταναλωτές, μεταξύ αυτών και τα γενετικά τροποποιημένα. Α, να πω και δύο λόγια για την επιστήμη τώρα, γιατί λένε ότι αυτό είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο, κουλουπού κουλουπού. Οι επιστήμονες πολλές φορές βλέπουν είτε αυτό που θέλουν να δουν ή αυτό τους είπαν ότι πρέπει να δουν. Αγνοούν λοιπόν κάποιες παραμέτρους. Στα γενετικά τροποποιημένα, κανείς σήμερα δεν μπορεί να πει τι μακροχρόνιες επιπτώσεις θα έχει η ο συσχετισμός γενετικά τροποποιημένου φυτού και φυτού που δεν έχει τροποποιηθεί γενετικά γιατί δεν έχουμε επαρκή στοιχεία. Γι' αυτό πρέπει να επιτρέψουμε να υπάρχουν και κάποιες αμφιβολίες ακόμα και όταν ε, το λόγο τον έχει η επιστήμη. Τελευταία παρατηρήση. Η μητέρα μου είναι 94 χρονών. Βλέπω ότι παίρνει του κόσμου τα φάρμακα κάθε μέρα. Πουθενά δεν μπορείς να διαβάσεις τι επιπτώσεις έχει το ότι παίρνει όλα τα, τα αυτά χάπια μαζί, γιατί κανείς δεν το μελέτησε. Τελευταία ερώτηση. Loving. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν είναι τόσο πολύ ερώτηση, αλλά περισσότερο σχόλιο σε μια προηγούμενη ερώτηση ενός συναδέλφου για το ότι δηλαδή ε, πλένουν τα κοτόπουλα με χλωρίνη κτλ. Εγώ ως λύση το βλέπω τελείως λάθος. Εγώ προέρχομαι από τη Σουηδία και καταφέραμε μέσω σωστής ε, κτηνοτροφίας αλλά και ε, σωστών νόμων ευημερία για τα ζώα καταφέραμε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο του σαλμονέλας πολύ πολύ πια περιθωριακές περιπτώσεις ε, εμφανίζονται και αμέσως εξαφανίζονται. Η εξάπλωση δηλαδή από τα ζώα στην Σουηδία είναι ανύπαρκτη και επίσης έχουμε τη χαμηλότερη ε, χρήση ιατρικών αντιβιωτικών στην Ευρώπη. Η Δανία χρησιμοποιεί τρεις φορές περισσότερα από τη Σουηδία, η Γερμανία 16 φορές και η Κύπρος 60 φορές περισσότερα αντιβιωτικά. Και αυτό γιατί, γιατί επιτρέπουμε με περισσότερο χώρο να έχουν τα ζώα, προβλέπουμε μάλλον, να έχουν περισσότερο χώρο τα ζώα και δεν ε, μεταδίδονται οι αρρώστιες τόσο εύκολα όσο όταν είναι στριμωγμένα σε περιορισμένους χώρους. Παρακαλώ λοιπόν καλύτερα δείτε ε, πώς θα κάνουμε εμείς στη Σουηδία. Ε, για να δείτε ε, ότι υπάρχουν τρόποι για να μην χρησιμοποιούνται τα αντιβιωτικά στα ζώα. Μάλιστα, έχουμε ενδιαφέρουσε ερωτήσεις. Έχετε τώρα εσείς την ευκαιρία να αντιδράσετε και να απαντήσετε. Μάλιστα. Πολλές καλές ερωτήσεις και κάποιες ε, διστάζω κάπως να τις απαντήσω γιατί νομίζω πως είναι πολιτικής φύσης και ίσως είναι καλύτερα κάποια από αυτά τα θέματα να τα συζητήσετε στην Επιτροπή σας. Ε αλλά εν πάση περιπτώσει θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Για την TTIP και την ασφάλεια των τροφίμων. Για μένα το πραγματικά σημαντικό θέμα εδώ για την ασφάλεια των τροφίμων και την TTIP, γιατί έχει πολλά μέσα, ξέρετε, πολλοί φόβοι εκφράζονται, ε, πολλοί κόσμος λέει ότι ε, ναι, θα προστατεύσουμε ψηλά πρότυπα ασφαλείας κτλ και νομίζω ότι από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, υποπαλλήλων και εδώ παντός Ευρωπαίου πολίτης. Αυτό που θέλουμε εδώ πραγματικά είναι η διαφάνεια, γιατί διαφορετικά μιλάμε για υποθέσεις και γενικότητες. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μπορούμε να δούμε τι θα κάνουμε με την ασφάλεια των τροφίμων και τη σχετική νομοθεσία, πώς θα λειτουργήσει και ε, Ποια θα είναι η πρόσβαση του κοινού. Επανεθνικοποίηση των γενετικά τροπομένων οργανισμών. Ε, αυτό είναι περίεργο και θα προσπαθήσω να καλύψω έτσι κάποιες ερωτήσεις. Υπάρχει αυτό το θέμα για το η ευελιξία δίνουμε στα κράτη-μέλη και το δούμε και αλλού σε άλλες πολιτικές όπως η κοινή γεωρική πολιτική, το πόσο, πόσο θα διατηρηθεί εντός της ε, ενιαίας αγοράς και πόσο όχι, πόσα μπορούμε να επανεθνικοποιήσουμε, γιατί η επανεθνικοποίηση είναι ενάντια στις αρχές της κοινή αγοράς και της Ένωσης. Νομίζω πως ε, υπάρχουν πολλά θέματα λοιπόν για τους γενικά τροποποιημένους οργανισμούς και ότι όταν υπάρχει τέτοια περίπτωση όπου 19 χώρες λένε όχι και το ευρύ κοινό επίση είναι πολύ ε, διστακτικό, τότε μάλλον κάτι πρέπει να μας κάνει να το σκεφτούμε περισσότερο. Αλλά είναι πολιτική φύση αυτή η συζήτηση και φαντάζομαι πως θα την ε, ε, κάνετε εδώ αυτή τη συζήτηση. Απλά θέλω να επανέλθω σε αυτή την ιδέα της επιστήμης, γιατί πρέπει να δούμε ναι, τις επιστημονικές αποδείξεις αλλά και άλλες πτυχές γιατί όταν μιλάμε για επιστήμη είμαστε ακαδημαϊκοί και έχουμε μια τάση να μιλάμε γενικά για τις ε, ιατρικές επιστήμες ή για τις φυσικές επιστήμες αλλά όχι αρκετά για τις κοινωνικές επιστήμες. Τώρα, το πλήσιμο με τη χλωρίνη. Υπάρχουν διάφορες λύσεις για την ασφάλεια των τροφίμων. Καταρχήν είναι το πολιτική απόφαση στην Ένωση να χρησιμοποιηθεί η προσέγγιση που ακολουθείται και αυτό για διάφορους λόγους. Υπάρχουν καλά παραδείγματα και για το κάμπυλο βακτηρίδιο αλλά και για τη σαλμονέλα όπου μπορούμε σχεδόν στην ουσία να τα εξαλείψουμε κάνοντας αλλαγές στην παραγωγή. Και υπάρχουν και οικονομικές εκτιμήσεις που έχουν νόημα σε ζεστό χρήμα, δολάρια και ευρώ. Ξεκονομείς δηλαδή χρήματα εφαρμόζοντας αυτά τα προγράμματα. Τώρα, γιατί βλέπουμε αυτές τις συνεχείς, τα συνεχή ξεσπάσματα. Για... Γιατί υπάρχουν διαφορές στο πώς εφαρμόζονται όλες αυτές οι πολιτικές στην Ένωση. Πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν την εφαρμογή και <laughs> να δούμε ποιες είναι οι καλύτερες πρακτικές για να, τα, να, να αυτά, αυτές, τα προβλήματα. Υπάρχουν τρόποι για να αλλάξουν οι παραγωγές μας. Γιατί εντάξει με τη χλωρίνη υπήρχαν σαφείς ενδείξεις ότι δεν θέλουμε τέτοιου είδους πολιτική ε, ασφάλεια των τροφίμων. Κύριε Πέτρελε, είπατε ότι ναι, θα πρέπει να είναι στο, ε, ε, στο προσκήνιο ο καταναλώτης. Ναι. Υπάρχουν πολιτικές όπου η δημόσια υγεία και η προστασία του καταναλωτή ήταν στον πυρήνα του, της προσπάθειας όπως το Λευκό Βιβλίο για την ασφάλεια στα τρόφιμα και η αντιμετώπιση της μεγάλης οικονομικής και υγειονομικής κρίσης της Τρελής Αγελάδας. Τώρα εξαρτάται από εσά αν θέλετε να παραμείνουν όλα αυτά κεντρικά θέματα. Και υπάρχουν ε, ζητήματα ε, μέσα στη διαδικασία REFIT που μπορεί να ε, θέσουν στο επίκεντρο τη συζήτηση σε αυτά τα ζητήματα. Ελπίζω να απάντησα στα ερωτήσεις σας ήταν μεγάλος ο κατάλογος και πρέπει να σας ομολογήσω ότι πολλές από αυτές πολύ δύσκολες μου φάνηκαν. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, ευχαριστώ όλους τους ομιλητές που ήρθαν σήμερα εδώ και που μοιραστήκατε μαζί μας τις ιδέες σας και μας δώσατε πολύτιμες πληροφορίες ε, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διάρκεια των ακροάσεών μας την επόμενη εβδομάδα, τις επόμενες δύο εβδομάδες μάλιστα. Ε, ήταν όλα αυτά λοιπόν πολύ ε, βοηθητικά θα μας βοηθήσουν πολύ για να δούμε πώς, με, τι μάτι θα δούμε τον υποψηφίου επίτροπες, πώς θα αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις προκλήσεις και τα προβλήματα που μας τονίσατε εσείς σήμερα. Ε, ε, τώρα ε, εδώ εμείς θα πρέπει να το, να το μελετήσουμε αυτό. Σας ευχαριστώ και πάλι λοιπόν για τη συμμετοχή και Εύχομαι και στους συναδέλφους καλή δουλειά για τις ακροάσεις και τέλος να ευχαριστήσω τη γραμματεία και σας συνάδελφοι που συνεργαστήκατε στην ε, πρώτη μου προεδρία <laughs> της Επιτροπής μας. Καλό σας απόγευμα.